στρατηγική θα επιβεβαιώσει αυτή την τάση και θα αυξήσει τη διαφάνεια, το, το διάλογο και περισσότερε διαβουλεύσει με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα Εθνικά Κοινοβούλια και την κοινωνία των πολιτών. Η στρατηγική είναι να εφαρμόσουμε αυτή τη στρατηγική και να λάβουμε υπόψη μα τη νέα πραγματικότητα. Γι' αυτό προετοιμάζουμε μια νέα ε, επικαιροποιημένη ε, εμπορική στρατηγική. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα. Γι' αυτό λοιπόν ήρθα εδώ για να ακούσω τι απόψει Φυσικά έχουμε έρθει σε επαφή με πολλούς από εσά, με τους συναδέλφους σας και πολλοί από εσά έχουν εμπλακεί στην όλη αυτή προσπάθεια. Έχουμε κάνει πάρα πολλά ταξιδεύοντας στα κράτη-μέλη, μιλώντας και ακούγοντας διάφορες Θα ήθελα όμως καταρχάς να σας πω κάποια πράγματα. Ε, ποιο είναι το νέο πλαίσιο και πώς ε, θέλουμε να αντιδράσουμε σε σχέση με αυτό. Η νέα εμπορική πολιτική έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, το εμπόριο πρέπει να είναι ατμομηχανή για τι ε, θέσει απασχόληση, ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων οικονομικών ε, ευκαιριών. Μία από τι 7 θέσει εργασία εξαρτάται ε, στι από τι εξαγωγέ στην Ευρώπη. Και συνήθω αυτέ οι δουλειέ είναι καλύτερα αμοιβόμενε. στο μέλλον, το 90% τη παγκόσμια ανάπτυξη θα προέρχεται από περιοχέ εκτό Ευρώπη. Άρα θα πρέπει το εμπόριο να μας βοηθήσει να, πετύχουμε αυτή την ανάπτυξη η Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου, ας πούμε, με, Βόρεια, με την Νότια Κορέα, ε, μπήκε ε, σε εφαρμογή το 2011 και αυξήθηκαν οι εξαγωγές μας στη χώρα αυτή κατά 35%. Αυτό που άλλαξε σήμερα είναι ότι οι οικονομία σήμερα είναι πολύ πιο στενά συνδεδεμένες από ό,τι παλιότερα και αυτό είναι το δεύτερο στοιχείο της εμπορικής μας Οι εμπορικές ροές ε, αγαθών και υπηρεσιών ε, παράγουν το 32% του παγκόσμιου ΑΕΠ και πολλές από τις εισαγωγές μας είναι ε, πρώτε και τα λοιπά, τα χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε προϊόντα που τα εξάγουμε μετά. Για να μπορέσουν λοιπόν οι εταιρείε μας να μετακινήσουν τα τελικά προϊόντα, θα πρέπει να μπορούν να παίρνουν τις πρώτε ύλε, εξαρτήματα κτλ. Ε, οι μεταφορές ε, το λιανεμπόριο είναι πολύ σημαντική τομή. Θα πρέπει να μπορούμε να δίνουμε υπηρεσίες, να διευκολύνουμε την ε, μεταφορά ανθρώπων, ε, τεχνικών, ε, μηχανικών κτλ. Παρόχων υπηρεσιών. Εδώ πάρα πολλά μπορούμε να κάνουμε για τις υπηρεσίες, που είναι το 40% της αξίας που προσθέτουμε στις ευρωπαϊκές εξαγωγές. Η μείωση των φραγμών εκτός θα είναι πολύ σημαντικό τα επόμενα χρόνια το να ανοίξουμε τα σύνορα, να, ανοίξουμε την, να αυξήσουμε την κινητικότητα. Είναι βασικό εργαλείο για να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα. Τρίτο στοιχείο της εμπορικής πολιτικής είναι ένα νέο πολιτικό περιβάλλον. Κάποιε από αυτέ τι αλλαγέ προέρχονται από μια έντονη συζήτηση που έχουμε για την ε, TTIP ε, με του ε, διατλαντικού εταίρους μα. Αυτή η στρατηγική εμπορική δεν αφορά μόνο το TTIP, αλλά έχουμε μάθει κάποια πράγματα από τη συζήτηση που έχουμε κάνει ειδικά σε διαφορά τη διαφάνεια και την ανάγκη να εξηγήσουμε και να δείξουμε στοιχεία, νούμερα, ε, για να, δούμε, να δείξουμε στον κόσμο τι κάνουν αυτέ οι διαπραγματεύσει. Οι καταναλωτέ δεν ζητάνε σήμερα μόνο χαμηλότερε τιμέ. Οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ θέλουν για να μάθουν πώ γίνεται το προϊόν που αγοράζουν, αν γίνεται ε, με μέσα σε αξιοπρεπεί συνθήκε, αν ε, οι εργάτε πληρώνονται, εάν ε, σέβονται βασικά κοινωνικά και περιβαλλοντικά δικαιώματα. Οι καταναλωτές πρέπει να ξέρουν για να επιλέγουν με τα λόγου γνώσεως και η εμπορική πολιτική πρέπει να απαντάει σε αυτές τις ανησυχίες. Όλο και περισσότεροι καταναλωτές πλέον είναι διατεθειμένοι να πλούσουν περισσότερα για προϊόντα δίκαιου εμπορίου. Θέλουμε να λάβουμε υπόψη μας αυτές τις αξίες. Ε, ανθρώπινα δικαιώματα, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει ότι αυτές οι αξίες θα υποστηρίζουν την ε, ευρύτερη εξωτερική ε, πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την πολιτική γειτονία. Περιμένω λοιπόν τις απόψει για το πώς θα τα προσεγγίσουμε όλα αυτά και να σα δώσω κάποιες από τι ιδέες μας. Πρώτον, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η εμπορική πολιτική είναι αποτελεσματική σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε νέα είδη εμπορικών φραγμών. Θα πρέπει να ανοίξουμε τι ε, υπηρεσίε. Ε, ζούμε στην ψηφιακή εποχή και αυτή έχει παγκόσμιο χαρακτήρα το άνοιγμα της ευρωπαϊκής αγοράς θα πρέπει να διατηρηθεί και να αναπτυχθεί περαιτέρω, ειδικά στην ψηφιακή οικονομία, ούτως ώστε οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις να έχουν ε, πρόσβαση στην ε, παγκόσμια αγορά, με προστασία βέβαια των ε, προσωπικών δεδομένων. Ε, αυτή η αγορά, η ψηφιακή αγορά, αξίζει σήμερα παγκόσμια πάνω από 12-3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις επιχειρήσεις. Μόνο λίγες από αυτές εξάγουν όμως πέρα από τα σύνορά μας. Ε, έχουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση για να τις βοηθήσουμε στις διαπραγματεύσεις στη ΤΥΠ και βλέπουμε πώς μπορούμε να τις λάβουμε υπόψη μας και σε άλλες διαπραγματεύσεις. Μια πιο αποτελεσματική πολιτική σημαίνει νέα εστίαση στην εφαρμογή των εμπορικών συμφωνιών. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τα ωφέλη των συμφωνιών φτάνουν όντως στους καταναλωτές, τις εταιρείε και τους εργαζόμενους. Και για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να έχουμε στενή εταιρική σχέση εμείς οι Κομισιόν με τα κράτη-μέλη που ελέγχουν την ε, πρόθεση των επενδύσεων. Και ελπίζουμε το Κοινοβούλιο να μας υποστηρίξει και εδώ. Ιδίω ό,τι αφορά τις, α, ε, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Δεύτερο στόχο, η νέα εμπορική στρατηγική ε, καθιστά το εμπόριο πιο υπεύθυνο. Θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να υλοποιήσουμε την εντολή μα, να προωθήσουμε τι ευρωπαϊκέ αξίε όλο τον κόσμο. Και αυτό ξεκινά με τη διαδικασία. Η δημοκρατία είναι ίσω η πιο θεμελιώδη αξία και έχει αμφισβητηθεί ε, μερικές φορές στα πλαίσια του εμπορίου. Ε, θα πρέπει να είμαστε πιο διαφανείς. Έχουμε ανοίξει επομένως την ε, Διατλαντική ε, Επενδυτική Συμφωνία και τη Συμφωνία για τις Υπηρεσίες. Και στις δύο αυτές διαπραγματεύσεις έχουμε βάλει στοιχεία online. Θα επεκτείνουμε αυτές τις πρακτικές και σε όλες τις άλλες διαπραγματεύσεις. Το να ξεπεράσουμε πέρα τώρα της διαδικασίας υπάρχουν οι κανόνες, προστασία των καταναλωτών, των περιβάλλων που ενσωματώνουν αυτές τις αξίες. Τα υψηλά μας πρότυπα δείχνουν ότι δίνουμε μεγάλη σημασία στο σεβασμό της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης ζωής και των ανθρωπίνων ελευθεριών. Έχουμε μία ανακοίνωση που δείχνει ξεκάθαρα ότι η κανονιστική συνεργασία δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μειώσει την προστασία. Για τις επενδύσεις, όπως ξέρετε, έχω προτείνει μια βαθιά μεταρρύθμιση στο σύστημα ε, και τη δημιουργία νέων, ε, ενός νέου επενδυτικού δικαστηρίου. Θα αναπτύξουμε περαιτέρω ε, αυτές τις ιδέες στην ανακοινώση για το εμπόριο. Η ακεραιότητα και στη διακυβέρνηση είναι βασική ευρωπαϊκή αξία. Αυτό με απασχολούσε όταν ήμουν επίτροπος εσωτερικών υποθέσεων. Το να καταπολεμήσω δηλαδή τη διαφθορά, Φερρυπίν. Είναι πολύ σημαντικό και στην ανακοίνωση θα λέμε πώ θα ε, το εξασφαλίσουμε αυτό με καλύτερε κρατικέ προπηρεσίε, διατάξει κατά τη διαφθορά σε όλε επίση τι εμπορικέ μα συμφωνίε. Επιπλέον, ε, βιώσιμη ανάπτυξη. Αυτό είναι ένα τομέα ε, όπου θα πρέπει να συνεχίσουμε να δείχνουμε ηγετικό ρόλο. Θα πρέπει και άλλε χώρε, ειδικά οι αναδυόμενε χώρε, να μα ακολουθήσουν. Θα πρέπει να δώσουμε νέε οικονομικέ ευκαιρίε, στους πιο φτωχού και θέλουμε να έχουμε ασφαλείς και αξιοπρεπείς συνθήκε εργασία και καθαρό περιβάλλον. Η ανακοίνωση θα πρέπει να προωθήσει την υπεύθυνη στρατηγική πάροχή υπηρεσιών και αγαθών και θα πρέπει να υποστηρίξουμε περισσότερο ε, το κίνημα δίκαιου εμπορίου και να υποστηρίζουμε τη δουλειά που κάνουν πολλές πόλεις και πολλοί μικιό. Διατάξεις για βιώσιμο περιβάλλον θα πρέπει να είναι ο κανόνα και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τι διατάξει των Συμφωνίων Ελευθερωμπορίου, τόσο ώστε να βοηθήσουμε και του εταίρου μα να προχωρήσουμε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι την ανακοίνωση, μέχρι να δημοσιευθεί, για να λάβουμε δράση, για να υποστηρίξουμε τι λιγότερο ανεπτυγμένε χώρε. Ζήτησαν ε, μία εξαίρεση από το κανόνα του ΠΟΕ για την πρόσβαση στο, στα φάρμακα σε ό,τι αφορά τις, μη λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες. Πέτυχαν αυτήν την εξαίρεση. Επίσης, στα αιτήματα που έχουν κάνει ΜΚΙΟ για το θέμα αυτό, απαντώ θετικά. Ο στόχος μου είναι να επικαιροποιήσω την διαπραγματευτική μου ατζέντα. Ε, εμείς θα πρέπει να υπερασπιστούμε το πολυμερές σύστημα σε, ένα κόσμο όπου πολλαπλασιάζονται οι διμερείς ε, συμφωνίες. Γιατί ο, ο υπομελής είναι και αξία και υπάρχει και συνθήκη, αλλά και είναι η καλύτερη απόκριση σε μια πακοσμιοποιημένη αλυσίδα αξιών. Είναι πολύ πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε τέτοιου τύπου συμφωνίες από διάφορες διμερείς συμφωνίες. Αυτό σημαίνει θα πρέπει το Ναϊρόμπι το Δεκέμβριο να τελεσφορήσουν οι διαδικασίες. Αλλά κοιτάμε και πιο πέρα. Βασικό στοιχείο και η βασική πρόκληση της εμπορικής πολιτικής είναι να πλουστεύσουμε τον αριθμό των ε, διμερών συμφωνιών που δημιουργούμε. Θα πρέπει να διαπραγματευτούμε πιο, ανοιχτές, ε, ε, πιο ανοιχτά και να διαπραγματευόμαστε πολυμερώς. Θα μπορούσαμε, παραδείγματο χάρη, και άλλες χώρες να μπουν σε, στις ισχύουσες συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και στο TTIP όταν ολοκληρωθούν. Και επίση οι υπόλοιπε συνδυμένε συμφωνίε θα πρέπει να γίνουν πιο συμβατέ μεταξύ του. Επίσης έχουμε και κάποιες, ε, κάποια εστίαση στην, ε, σε γεωγραφικές ζώνες. Ε, Ασία, ε, ειρηνικός. Πιο βαθιά σχέση με την Κίνα θα πρέπει να προχωρήσουμε τους ε, εταίρους ΑΣΕΑΝ και να έχουμε επενδυτικέ συμφωνίε με άλλε χώρε Ασία. Επίση με χώρε όπω Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία. Πιο βαθιά σχέσει. Έχουμε τόσε κοινέ αξίε και αξίζει να το κάνουμε. Η οικονομική συμφωνία έχει μια, δώσει μια νέα δυναμική στη... και έχει εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε δύο υπήρους εμάς και στην... Και μπορούμε να προχωρήσουμε και με τις επενδύσεις στα πλαίσια της Συμφωνίας Ε, και μπορούμε λοιπόν να έχουμε καλύτερη συνεργασία ανάμεσα σε εμά και στη Λατινική Αμερική. Μπορούμε πολύ γρήγορα να αρχίσουμε να εξυγχρονίσουμε τη συμφωνία μας με το Μεξικό και τη Χιλή και να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία ξεκινώντας με τις διαπραγματεύσεις για βαθιά ε, συμφωνία ελευθέρου εμπορίου με το Μαρόκο και ελπίζουμε να ξεκινήσουμε και διαπραγματεύσεις με την Τινησία. Για να τα κάνουμε όλα αυτά θα πρέπει να συνεργαστούμε από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Νομίζω ότι έχουμε και αποτελεσματικούς αλλά και φάνταστους τρόπους για να συνεργαστούμε. Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά όταν το κάνουμε ε, τα αποτελέσματα πάντα είναι πολύ καλά για τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Για να εξυγχρονίσουμε την εμπορική μας πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να είναι αποτελεσματική, για να είναι υπεύθυνη και για να είναι στοχευμένοι οι στόχοι μα ε, για να χρησιμοποιήσουμε του σωστού εταίρου. Πρέπει να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε και πρέπει να έχουμε περισσότερη συνεργασία. ιδέε ο ζήλος σας, η απόψη σας και η σχέση και η επαφή που έχετε με τους ανθρώπους που προσωπείτε θα είναι σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία. Περιμένω λοιπόν τις σημερινές απόψεις και τις επόμενες μέρες και πιστεύω ότι θα έχουμε καλή συνεργασία. Περιμένω τώρα τις ερωτήσεις σας, Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Επίτροπε. Ξεκινάμε με τον πρώτο γύρο παρεμβάσεων των συντονιστών και θα ακολουθήσουν τα άλλα μέλη στο δεύτερο γύρο. Από το ΕΛΚ. Κύριος Κασπάρη, παρακαλώ. Μάλιστα. Αγαπητέ Επίτροπε, σας ευχαριστούμε πολύ αγαπητή Επίτροπε για την παρουσίασή σας και ευχαριστούμε που είσαστε εδώ. Θέλουμε πρώτα απ' όλα να συστήσουμε, να σας εκφράσουμε θερμές ευχαριστίες. Αυτά που είδαμε κατά τους πρώτους 7 μήνες της θητείας σας ως Επιτρόπου είναι μια πολύ καλή προσέγγιση, νέα προσέγγιση σε σχέση με τον προκατοχό σας και είμαστε ικανοποιημένοι διότι θέλετε, έχετε την βούληση να εμπλακείτε περισσότερο, να εμπλέξετε περισσότερο τους πολίτες, να υπάρξει μεγαλύτερη διαφάνεια. Είδαμε τις πρώτες επιτυχίες κατά τον προηγούμενο μήνα και σας υποστηρίζουμε και μελλοντικά στη δράση σας αυτή. Θα αλλάξω τώρα και θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα τα γερμανικά. Το πρώτο θέμα που με ενδιαφέρει είναι η πολυμερής προσέγγιση του Διεθνούς Οργανισμού Εμπορίου. Είχαμε κάποιες δυσκολίες να κλείσουμε το πακέτο του Μπάλι και είχαμε δυσκολίες επικύρωσης. Και τώρα η ερώτησή μου, βλέπετε κάποια ευκαιρία στην Κένια τώρα στη συνέχεια σε κάποιο από τα συγκεκριμένα πακέτα να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες ή να κάνουμε τουλάχιστον ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός. Και αν ναι, Ποια θέμα, σε ποια θέματα θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτό. Δεύτερον, TTIP, η Συμφωνία Επενδύσεων και Εμπορίου με τη ΣΥΠΑ. Αυτή την εβδομάδα θα γίνουν διαπραγματεύσεις στις Βρυξέλλες. Ερώτησή μου, τους εκπροσώπους από πλευράς ε, τον είπα, θα τους επισημάνετε ότι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη εβδομάδα με μεγάλη πλειοψηφία αποφάσαμε σχετικά το τι πρέπει να γίνει. Καλό μήνυμα θα ήταν να συζητήσετε με τους Αμερικανούς και να ληφθούν υπόψη οι προκλήσεις και οι δυσκολίες και οι στοχοθετήσεις που έχουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τρίτον, το ερώτημα πότε συγκεκριμένα θα έχουμε το κείμενο ώστε με τη διαδικασία επικύρωσης να ξεκινήσουμε επίσημα. Τέταρτο, Βλέπετε κάποια πιθανότητα, κάποια ευκαιρία κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Είμαι πολύ προσεκτικός στη διατύπωση. Τις συμφωνίες με την Κίνα, Ταϊβάν, Βιετνάμ να τις ολοκληρώσουμε από κοινού λοιπόν Βιετνάμ, Ταϊβάν, Ιαπωνία, Κίνα, τα αναφέρω αυτά τα κράτη. Βλέπετε κάποια ευκαιρία να ολοκληρωθούν στη θητεία σας αυτά τα τέσσερα θέματα αυτών των τεσσάρων συμφωνιών. Και πέμπτο θέμα, συνεργασία για παράδειγμα με τους συναδέλφους σας όσον αφορά φόρους και δασμούς. Έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει αυτά τα θέματα. Ξέρουμε ότι υπάρχει εδώ, εδώ θέμα της αρμοδιότητας So, ähm, stört uns weiterreden. Δεν μας ενοχλεί καθόλου, μπορούμε να συζητήσουμε και να ακούμε ένα τον άλλον. Το θέμα της, ε, των ε, δασμών ε, στα εξωτερικά μας σύνορα με τα κράτη-μέλη βλέπετε κάποια ευκαιρία να συζητηθεί και έχουμε και την αποστολή πριν από λίγες εβδομάδες στην Ιταλία όπου είδαμε πόσο διαφορετικά αντιμετωπίζονται από τα 28 κράτη-μέλη και τις υπηρεσίες τους τα θέματα των τελωνίων και εντωμεταξύ έχουμε και ανταγωνι... θέματα ανταγωνισμού ε, και τα θέματα ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών και την εισαγωγή ε, εμπορευμάτων υπό αυτή την πτυχή. Βλέπετε κάποια πιθανότητα να μπορέσετε να προχωρήσετε στα θέματα αυτά με τα κράτη-μέλη κατά τη διάρκεια της θητείας σας. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια για τους σοσιαλδημοκράτες έχετε εσείς τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να δω τις σημειώσεις μου βέβαια με στο σκοτάδι. τι να κάνουμε. Και εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω την Επίτροπο για το έγγραφο αυτό. Είναι σημαντικό. Να πω ότι η πρώτη έκκληση προς την Επίτροπο είναι ότι αυτό το έγγραφο θα πρέπει να έχει πολλές φιλοδοξίες. Θα πρέπει να είναι όσο πιο φιλόδοξο γίνεται. Δεν πρέπει να είναι ένα έγγραφο που θα αφορά αυτούς που ασχολούνται με το εμπόριο ή τους εργοδότες. Γιατί στις ε, εφημερίδες που διαβάσαμε είδαμε ότι υπάρχει μια εστίαση στο εμπόριο. Όμως το εμπόριο είναι ένας μοχλός για να επιλύσουμε διάφορα άλλα θέματα που είναι ανοιχτά, που ίσως τα τελευταία χρόνια δεν καταφέραμε να επιλύσουμε. Ίσως γιατί είχαμε τα μάτια μας πολύ στραμμένα στο εσωτερικό μας. Υπήρχε ένα είδου στρουφοκαμιλισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτό το έγγραφο, με αυτή τη νέα στρατηγική, νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μια συνεισφορά. Α. Ως Ευρώπη στον κόσμο. Και να επιλύσουμε και κάποια προβλήματα τα οποία υπάρχουν και επανέρχονται και που τα είδαμε και αυτές τις τελευταίες μέρες έντονων διαπραγματεύσεων. Καταρχάς, τι σημαίνει ε, μια νέα δημοκρατία στα πλαίσια της νέας παγκοσμιοποίησης. Πώς εμείς, ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, μπορούμε να απαντήσουμε σε τέτοιου τύπου ερωτήματα. Νομίζω ότι μια τέτοια στρατηγική ε, πρέπει να υπάρχει. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτούς τους προβληματισμούς. Αυτό το έγγραφο μπορεί να γίνει ένα μανιφέστο του τι σημαίνει η νέα Ευρώπη και γιατί πρέπει να δρομολογήσουμε αυτό το νέο project. Και η εμπορική πολιτική είναι ένα από τα κλειδιά για να ξεκλειδώσουν αυτό το παζλ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε τέτοιου τύπου γενικό προβληματισμό. Για να πάμε τώρα σε επιμέρους θέματα. Πρώτον, εκτιμώ πολύ την επιμονή που δείχνεται για τη διαφάνεια στις διαπραγματεύσεις. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε ακόμα ένα βήμα. Υπάρχει μια τέτοια έλλειψη εμπιστοσύνης, μια δυσπιστία απέναντι στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, που δεν νομίζω ότι αρκεί να μιλήσουμε απλώς για διαφάνεια και να επικοινωνούμε απλώς. Νομίζω ότι θα πρέπει να αλλάξουμε άρδιν. Πρέπει να γίνει μια τεράστια προσπάθεια και να υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα στους πολίτες και στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εδώ είναι σημαντικός. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε απόλυτη διάθεση να βρούμε τους πιο καινοτόμους, τους πιο νέους τρόπους για να ανακτηθεί λιγάκι η χαμένη εμπιστοσύνη. Τώρα, για πιο συγκεκριμένα ακόμα θέματα, νομίζω είναι σημαντικό, όπως τονίσατε κι εσείς, να συνδέσουμε στενά την πολιτική που προωθούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με το Digital Single Market, την ψηφιακή ενιαία αγορά, γιατί από όλες τις πολιτικές αυτή είναι η, πιο, η πλέον συνδεδεμένη και η πιο συναφής με την εμπορική πολιτική. Θα πρέπει να δούμε πώς θα συνδεθούν αυτές οι δύο πολιτικές λοιπόν. Η πολιτική, η εμπορική με την ψηφιακή ενιαία αγορά. Θα ήθελα να μου πείτε κάποια πράγματα για την Κίνα τώρα. Για την διάσκεψη του Παρισιού που θα γίνει στο τέλος του 2015 και στα ντοσιέ που θα φτάσουν στο τραπέζι μας και για τις α, ε, πολυμερείς συμφωνίες, η Κίνα τι ρόλο μπορεί να παίξει. Ευχαριστώ. Αγαπητοί συναδελφοί, άφησα να μακρηγορήσουν κάπως οι πρόσωποι των μεγάλων ομάδων. Τώρα, οι υπόλοιποι παρακαλώ να είσαστε το δυνατόν συντομότεροι. ECR, Τέμπελ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, όπως γνωρίζετε είμαι εισηγητής για την Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου ΕΕ Ινδίας. Καλωσορίζω πολύ την συνάντηση σε σχέση με τα τέλη Αυγούστου. Διαρωτώ με υπάρχουν και κάποια άλλα σημεία πρόοδου που μπορείτε να αναφέρετε σχετικά από πλευράς αντιπροσωπείας ΕΕ Ινδίας. Είχαμε εκπροσώπους ε, που ε, είχαν προσέλθει και ε, υπήρχε υπήρχαν πολλές ε, ανησυχίες ε, για τα θέματα της ε, γεωργίας. Διερωτώ με, θα θέλατε να το σχολιάσετε αυτό. Και τέλος, μια μεγάλη ανησυχία για τα θέματα πολιτικής σας, τα οποία επικεντρωνόμαστε όσον αφορά πολιτικούς στόχους. Την αηφοροανάπτυξη, για παράδειγμα, δικαιώματα του ανθρώπου και τα συναφή δημιουργούνται προβλήματα σε σχέση με αυτά με, την, το ελεύθερο εμπόριο με την Ινδία και υπάρχουν και θέματα με την Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Θα μπορούσατε να τα σχολιάσετε. Θα συνεχίσουμε ε, αυτή την πορεία διότι ε, σε σχέση με το ευρώ για παράδειγμα και το να δούμε πού θα ε, ολοκληρωθούν και πώς θα τελειώσουν τα πράγματα πρέπει να δούμε σε σχέση με το ελεύθερο εμπόριο ποιες προοπτικές υπάρχουν. Εσείς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Για την έκφραση των, των ιδεών σας εδώ για το ελεύθερο εμπόριο. Έχουμε αρκετές ευκαιρίες τελευταία να κάνουμε τέτοιες ανταλλαγές απόψεων και εκτιμώ ιδιαίτερα το ότι συμφωνείτε και εσείς τονίσατε τις αξίες και τις αρχές στις οποίες βασίζεται η Ένωσή μας και που πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε κάθε εμπορική μας συμφωνία. Είναι επίσης προκλητικό αλλά και ενδιαφέρον να δούμε πώς θα το εφαρμόσει αυτή την πρόκληση η Ένωση. Σε πανενωσιακό επίπεδο τα λέμε πρόσφατα μόνο τα εμπορικά. Παρά την επικουρικότητα. Και θα ήθελα να μου πείτε λίγο ευρύτερα πώς βλέπετε εσείς ε, την πολιτικοποίηση του παγκοσμιοποιημένου εμπορίου. Ότι έχει πολιτικοποιηθεί είναι φανερό, το βλέπουμε στις σχέσεις μας με τη Ρωσία αλλά και τον κόσμο που αλλάζει λόγω της ψηφιοποίησης των αναδειωμένων οικονομιών αλλά και την πίεση που υφίστανται οι εμπορικές σχέσεις και με τα Βεβαίως αναφέρατε ότι 90% της παγκόσμιας ανάπτυξης θα σημειωθεί εκτός Ένωσης. Ως λοιπόν εμπορικές και εξαγωγικές οικονομίες από εκεί βγάζουμε εμείς τα κέρδη μας αλλά με τι κανόνες. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους και θα ήθελα να μας πείτε πώς θα μπορέσουμε να φτάσουμε να αποφύγουμε την εξουδετέρωση, την πλήρη εξουδετέρωση μας. Θέλουμε η ανάπτυξη να υπάρξει ακόμη και αν καμιά φορά κλείνουμε τα μάτια σε αρχές και τρόπους που λέμε ότι είναι η βάση της κοινωνίας μας. Μπορούμε λοιπόν να ενδυναμώσουμε το σύστημα του σεβασμού των κανόνων, με τα ανθρώπινα δικαιώματα, με, το, με μέτρα καταπολέμησης του ντάμπινγκ ή το παράδειγμα της Κίνας. Το θέμα είναι θέλουμε ή όχι να επιβάλλουμε ή να επιμείνουμε στους κανόνες και τις ιδέες που θεωρούμε ότι πιστεύουμε αλλά που καμιά φορά στην πράξη δεν το βλέπουμε. Α πούμε αν διαπιστώσουμε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων τι θα κάνουμε αν δούμε περίπτωση dumping για πολιτικούς λόγους θα πάρουμε μέτρα ή όχι και χαίρομαι που αναφέρατε επίσης την έμφαση που δίνει η Επιτροπή για άλλα μέρη του κόσμου όπως την Αφρική πρέπει φυσικά η πολιτική γειτονία να είναι από τα κύρια θέματα της εμπορικής μας πολιτικής. Θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω και για την Δημησία και την Ουκρανία, όπου υπάρχει και εκεί ένα θέμα πολιτικοποίησης του εμπορίου, γιατί η Ρωσία πιέζει και την Ένωση και την Ουκρανία για να αλλάξουν οι συσχετισμοί και οι κανόνες εκεί του εμπορίου. Αυτό κυρίως λοιπόν η πολιτικοποίηση και πώς θα ε, ισχυροποιήσουμε το σύστημα σεβασμού των κανόνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ Επίτροπε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτή τη νέα προσέγγιση που υιοθετήσατε σε μια διαρκή και σε βάθος ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση με την ε, Επιτροπή Παγκοσμίου Εμπορίου δίνει θετικές προοπτικές στο να επικεντρωθούμε στα πιο φλέγοντα και σημαντικά θέματα που έχουμε ενώπιόν μας. Και καθώς ε, συζητάμε αυτά τα θέματα πολύ συγκεκριμένα υπό πολύ σημαντική συγκυρία με την κρίση του ευρώ και την δημοσιονομική κρίση και τις εξελίξεις, πρέπει να γίνει κατανοητό ότι εμπορικές πολιτικές συνάδουν με τις οικονομικές πολιτικές όχι μόνο με τα θέματα τα νομισματικά και όχι μόνο με την αποστολή εμπορευμάτων από ένα σημείο σε άλλο, αλλά πώς και με, πού μπορεί να συνεισφέρει το εμπόριο στην αηφόρο ανάπτυξη. Και αυτό αληθεύει και για όλα τα κράτη-μέλη και για τις προσπάθειές τους. Και έτσι λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο, με εξέπληξε το γεγονός ότι δεν κάνατε λόγο για την παγκοσμιοποιημένη Ευρώπη, Global Europe, γιατί σε σχέση με την παλαιά στρατηγική αυτό ήταν ένα κύριο στοιχείο και το βρήκα πολύ πιο ενθαρρυντικό ότι εσείς κάνατε λόγο για τις τομεακές πολιτικές του εμπορίου την ανάγκη να προσθεθούν στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι κλιματικές αλλαγές, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι ευκαιρίες ε, του να αντιμετωπιστεί η φτώχεια, να εκριζωθεί η φτώχεια και θα ήθελα εδώ να προσθέσω και την ερώτησή μου προς εμάς Επίτροπε εδώ. Να σας πω ότι αν ακόμα και πριν από τη συνθήκη της Λισαβόνας κατά το παρελθόν όταν είχαμε αρμοδιότητα και κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών για διμερείς εμπορικές συμφωνίες και στο όνομα της Ευρωπαϊκής ε, ε, Ένωσης δεν καταφέραμε να εκριζώσουμε την φτώχεια και δεν μπορέσαμε να προχωρήσουμε όπως έπρεπε σε σχέση με τα όσα συνέβησαν πριν από 10 ή 15 χρόνια. Και εδώ το πολυμερές σύστημα εμπορίου που πρέπει να καταστεί λειτουργικό προς όφελος των πολιτών. Το ερώτημα μου είναι πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή για το άμεσο μέλλον προσεχώς την ευκαιρία τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υποστηρίξουν την δική σας προσέγγιση για μια ευρωπαϊκή πολιτική για το εμπόριο όπως ε, εσείς την παρουσιάσατε και την προωθείτε και ευχαριστώ για την πρόσκληση καθένας και κάθε μια από μας να μπορεί να συμμετάσχει και όσον αφορά την περαιτέρω διατύπωση και προώθηση της ανακοίνωσής σας ώστε να υπάρξουν προτάσεις που θα ληφθούν υπόψη από πλευράς μας. Και η Ευρωπαϊκή ημέρα παγκοσμίου εμπορίου νομίζω ήταν ένα σωστό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση σχετικά. Και τέλος, ολοκληρώνοντας, αναφέρατε τις γεωγραφικές προκλήσεις. Διαρωτώ με, θα μπορούσατε να εξειδικεύσετε περισσότερο να αποσαφηνίσετε περισσότερο έναντι της Ανατολικής Ευρώπης και τις γειτονικές χώρες, τις χώρες γειτονίας προς την Ανατολική Ευρώπη και τις Κεντρασιατικές χώρες, τι γίνεται και τη Ρωσική Ομοσπονδία, πώς και πού μπορούμε εμείς να συνεργαστούμε με αυτές τις χώρες. Τι μπορούμε να κάνουμε, δίνοντας συνέχεια στο σημαντικό ζήτημα, πώς το εμπόριο μπορεί να συνεισφέρει να ξεπεράσουμε σειράξεις, ε, τριβές, ε, αντιπαραθέσεις κτλ. Και βλέπετε κάποια συνάφεια με τους άλλους πυλώνες στην ε, ευρωπαϊκή πολιτική εξωτερικής δράσης από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. <coughs> Κυρία Επίτροπε, μιλήσατε στην αρχή για τις συνεννοήσεις που είχατε με πολιτικές ομάδες Έγινε λόγος επίσης γενικά για επικοινωνία. Φαντάζομαι ότι με κλήρο τα κανονίσατε γιατί εμάς δεν μας ε, διαβουλεύτηκε κανείς για αυτό το θέμα. Οι συνάδελφοί μου θα επανέλθουν στο θέμα της στρατηγικής Σήμερα είμαι πολύ απογοητευμένος από την Ευρώπη. Νομίζω ότι ζούμε πολύ άσκημες ώρες στην Ένωση που μάλλον δεν είναι καν πια ένωση αλλά μία Ευρώπη εθνών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ποτέ μέχρι τώρα δεν είχε βασιστεί στον κινησμό και στα λογιστικά και στην ταπείνωση και νομίζω ότι ακόμη μια φορά, το ξαναλέω, για πρώτη φορά εδώ και 60 χρόνια παίχτηκε ως στίχημα η αποδόμηση ενός τμήματος της Ευρώπης. Με βάση αυτά που έγιναν στην Ελλάδα αλλά και γενικότερα για τα εμπορικά. Η Ελλάδα θα χρειαστεί και αυτή η εμπορική συνεργασία και οι εμπειρογνώμονες θα λένε πριν ακόμη αποφανθεί ο νομοθέτης αν μπορεί να αποφανθεί και πώς. Βέβαια όταν κανείς διαχειρίζεται ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που βασίζεται στη λιτότητα και την οικονομική ασφυξία η εμπορική πολιτική κατευθύνεται αναγκαστικά προς την εξέβρεση αγορών και σήμερα έχω σοκαριστεί παραπάνω από ό,τι συνήθως τρομερά που χρειάζεται να υπερασπιστώ μια Ευρωπαϊκή Ένωση που ξεχνάει την αλληλεγγύη, ξεχνάει την πολιτική βασίζεται σε διαιρέσεις μεταξύ χρεωστών και οφειλετών και νομίζω ότι αυτό δεν με καθυσχάζει καθόλου γιατί υπάρχουν κινήματα και τάσεις στην Ευρώπη που θα κερδίσουν τελικά και που τραβάν την Ευρώπη προς τα κάτω. Ευχαριστούμε κυρία Μπεγκίν. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε σήμερα στην Επιτροπή μας για να μας παρουσιάσετε τη μελλοντική εμπορική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μου συμβαίνει συχνά να σας απευθύνω το λόγο μιλώντας σας για την DTIP. Ε, χαίρομαι που αλλάζουμε και λίγο θέμα για μια φορά και δεν μιλάμε για τα ίδια και τα ίδια. Χαίρομαι που θα μιλήσουμε σήμερα για αυτό το θέμα. Εγώ πιστεύω στη σημασία του εμπορίου. Πιστεύω στη σημασία αυτής της Επιτροπής, γιατί το εμπόριο έχει το δυναμικό να επηρεάσει τη ζωή των ανθρώπων να επηρεάσει πράγματα και δεν πιστεύω στον προστατευτισμό ούτε στην, στον άκρατο εμπορικό ανταγωνισμό. Πιστεύω στη συνεργασία, στην αμοιβαία αναγνώριση των διαφορών μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στο εμπόριο. Το εμπόριο μας βοήθησε να ξεπεράσουμε τα σύνορά μας το παρελθόν μας βοήθησε να αναγεννηθούμε από τις τάχτες μας. Ακόμα και σήμερα μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε το εμπόριο για να βγούμε από την οικονομική κρίση. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα εμπόριο το οποίο θα βασίζεται σε κανόνες που θα, τα, θα τους εφαρμόζουν όλοι μας οι εμπορικοί εταίροι για να είναι πραγματικό αναπτυξιακό εργαλείο αυτό, όπως και εσείς είπατε. Για, και για να γίνει αυτό θα πρέπει να ξαναδούμε πώς λειτουργεί ο ΠΟΕ, η Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου, πώς κατηγοριοποιούνται οι χώρες στο εσωτερικό του, να δώσουμε περισσότερο χώρο σε πολυμερείς συμφωνίες κτλ. Θα πρέπει λοιπόν να ολοκληρώσουμε τον κύκλο της ε, Ντόχα, να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για το εμπόριο του Μπενιβέρντι, να υπάρχει πάντα ένα κεφάλαιο βιώσιμης ανάπτυξης, όχι μόνο σε διμερές αλλά και σε πολυμερές επίπεδο στο διμερές επίπεδο θα πρέπει να οργανωθούμε ούτως ώστε να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της TTIP στις ε, αγορές μας. Να αρχίσουμε να μιλάμε με χώρες που μπορούν να μας βοηθήσουν ούτως ώστε να έχουμε πρόσβαση σε άλλες αγορές οι οποίες αυτή τη στιγμή υπογράφουν το TTIP. Θα πρέπει να, να, να ξαναρχίσουμε τις συζητήσεις που έχουμε σταματήσει με την Ινδία, Φερρυπίν. Να ξεκινήσουμε από το θέμα επίλυσης του προβλήματος με τους δύο Ιταλούς που κρατάει η Ινδία στην επικράτειά της. Θα πρέπει να δούμε επίσης την προσέγγισή μας απέναντι στην Κίνα και η πολιτική των επιδοτήσεων θα πρέπει να σταματήσει. Ούτω ώστε να έχουμε όχι μόνο δίκαιη πρόσβαση στις αγορές, αλλά αύξηση και της παραγωγής μας. Νομίζω ότι με αυτές τις χώρες πρέπει να βρούμε μια συνεργασία. Όχι αντιπαράθεση, συνεργασία. Αλλά θα πρέπει να ξέρουμε ότι όλο και περισσότερο μαθαίνουν για το πώς θα επηρεάσουν τις διαδικασίες που τους επηρεάζει και χρησιμοποιούν τα στοιχεία που έχουν προς όφελός τους. Δεν θα πρέπει να αφαιθούμε και να νικηθούμε. Θα πρέπει να ζητήσω κάποιε διευκρινήσει για ένα θέμα το οποίο με απασχολεί τα μάλα, το made in, του ελέγχου και τι πιστοποίησει ποιότητα. Δεν είναι θέμα σημαία αυτό. Νομίζω ότι όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτε θα πρέπει να είναι σίγουροι ότι αυτό που καταναλώνουν και αγοράζουν παράγεται στην Ευρώπη ή οπουδήποτε αλλού και όπου και να παράγεται έχει κάποια, βασίζεται σε κάποια πρότυπα ασφάλειας και οι εταίροι μας θα πρέπει να αρθούν στο δικό μας ύψος και όχι εμείς να κατέχουμε στο δικό τους. Αυτό που είπε ο κ. Κάσπαρη, το θέμα των τελωνίων, πολύ σημαντικό. Ε, και έκανα μια επίσκεψη μαζί με τον κ. Φίσα στην ε, Γενέβη, συγγνώμη στη Γένοβα, ε, και πρέπει να ξαναδούμε τι ε, τελωνιακέ ε, πρακτικέ πραγματικά, ώστε να υπάρχουν τα ίδια επίπεδα προστασία σε όλα τα λιμάνια. Τελευταίο σημείο. Το εμπόριο, νομίζω, είναι ένα ωκεανό ευκαιριών για μα και για του εταίρου μα. Αλλά νομίζω, για να δράξουμε την ευκαιρία, θα πρέπει το σκάφο μα να είναι αξιόπλο. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τι εργαλεία δεν λειτουργήσαν στο παρελθόν, τι εργαλεία έχουμε αμυντικής φύσεως, τα οποία δεν χρησιμοποίησαμε καλά στο παρελθόν. Θα ήθελα περισσότερε εξηγήσει γι' αυτό. Ο κύριο Ραν τώρα παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Επίτροπε. Εγώ είμαι νεοφερμένος εδώ στην Επιτροπή σας και Μιλάω πάντοτε περισσότερο για τα γαλλικά συμφέροντα. Ε, μιλήσατε κυρία Επίτροπε για τους καταναλωτές, λες και οι Ευρωπαίοι πολίτες είναι εμπορεύματα με μόνο στόχο να γίνονται ελεύθερες συναλλαγές με τη Διατλαντική Συμφωνία. Θα ήθελα και εγώ να σας μιλήσω για το τι πιστεύουν οι Ευρωπαίοι γι' αυτό. Δύο δημοσκοπήσεις, μία παλιά, μία πιο πρόσφατη, δείχνουν ότι στη Γαλλία ιδίω υπάρχουν μεγάλες δυσκολίες για την καθημερινή ζωή των πολιτών και φοβούνται πάρα πολύ οι καταναλωτές το μέλλον. Η πρώτη δίσκη ότι κατά 70% οι Γάλλοι είναι κατά των ελευθερών συναλλαγών και ότι θέλουν προστατευτική πολιτική. Η δεύτερη δημοσκόπηση από το ΙΦΟΠ δεν αφορά μόνο τους Γάλλους αλλά και τους Ιταλούς, τους Ισπανούς, τους Γερμανούς φετινή είναι αυτή η δημοσκόπηση, η προηγούμενη ήταν του 11 και δείχνει ότι είναι πάντα οι πολίτες κατά των ελευθέρων συναλλαγών και προτιμούν τα πρότυπα που ίσχυαν πριν. Επομένως κυρία Επίτροπε, πώς δικαιολογείτε ότι εφαρμόζεται τόσο ακραία νεοφιλελεύθερα μέτρα ενώ οι πολίτες είναι κατά. Δυστυχώς Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πιο νεοφιλελεύθερη οντότητα του κόσμου, έχει το χαμηλότερο ρυθμό ανάπτυξης στον κόσμο. Και από πολύ καιρό. Η στρατηγική λοιπόν που μας προτείνεται είναι αποτυχία. Επομένως κυρία Επίτροπέ μου, τίθενται πολλά ερωτήματα εδώ. Η βιομηχανία και η γεωργία θα αποτελέσουν τα θύματα που θα σφαγούν εν ονόματι αυτής της ιδεολογίας ή θα επιλέξετε επιτέλους λύσεις που θα βοηθήσουν τους πολίτες μας. Χρειάζονται κανόνες, ναι. Και αν δεν υπάρχουν, αν δεν τους ξέρετε, μπορώ να σας αναφέρω δύο. Η μία για, την αμπελοϊνη, για το αμπελοϊνικό για τις αμπελοϊνικές δραστηριότητες. Υπάρχουν κανόνες για τα δικαιώματα εμφύτευσης και είδαμε ότι τα μπελοϊνικά είναι πολύ σημαντικό τμήμα της δραστηριότητας μας. Έπειτα οι γαλακτοκομικές ποσοστώσεις που απελευθερώθηκαν ήταν πλήρης αποτυχία. Και στη Γαλλία αρχίζει να φαίνεται αυτό, να γίνονται παντού διαδηλώσεις και σχεδόν εξέγερση. Καταλήγω λοιπόν κύριε Πρόεδρε απλώς ότι θελήσατε Ευρώπη των 28, ήδη ήταν πάρα πολλά τα μέλη. Τώρα κάνουμε συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών και με την Τινησία, το Μαρόκο, την Τουρκία, τη Μολδαβία και άλλες χώρες με τις ίδιες συνθήκες τάχα που ισχύουν στην Ένωση. Ως πού θα φτάσετε κυρία Επίτροπε. Ποια είναι τα συμφέροντα των Ευρωπαίων πολιτών μπροστά σε αυτή την κρυμμένη διεύρυνση. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί συνάδελφοι, οκτώ έχουν ζητήσει ακόμη τον λόγο. Παρακαλώ, ίσως ένα λεπτό ο καθένας. Όχι πιο πολύ. Να τηρήσουμε αυτό το όριο, ώστε να μπορέσουν όλοι να παρέμβουν. Ο κύριος Βαλένσα πρώτος, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για την Κίνα και την οικονομία και την αγορά της. Ίσως είναι μια πιθανή πυρητιδαποθήκη για την ευρωπαϊκή βιομηχανία και ελπίζω να το ξέρετε. Μια συγκεκριμένη ερώτηση λοιπόν. Χαίρομαστε που έχουμε χαμηλούς δασμούς, που είμαστε ανοιχτοί στις υπηρεσίες στις κρατικές προμήθειες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η πιο ανοιχτή και μεγαλύτερη αγορά στον κόσμο. Αν κοιτάτε όμως τις προοπτικές που έχουμε, αν θέλουμε να ανταγωνιστούμε την Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, Ρωσία, τις μεγάλες αυτές αγορές, νομίζω ότι οι ή εξαγωγής μας δυσκολεύονται να αντιδύσουν στην Κίνα και την Βραζιλία όλους ιδιαίτερος. Από την ανακοίνωσή σας και τις δηλώσεις σας ε, συνάγω ότι η λύση σε αυτό το πρόβλημα είναι περισσότερη απελευθέρωση του εμπορίου. Περισσότερες συμφωνίες, δηλαδή ελεύθερου εμπορίου, με το Μερκοσούρ, την Ινδία και επενδυτικές συμφωνίες ε, με την ε, Κίνα. Όλο καρότα τους δίνεται. Κάνα μπαστούνι δεν έχει. Θεωρείτε ότι το να κλείσουμε τις ευρωπαϊκές αγορές στις ε, κρατικές προμήθειες, ας πούμε, ή στις υπηρεσίες χωρών που δεν ανοίγουν τις αγορές στους δικούς μας παραγωγούς, δεν είναι μια λύση. Φυσικά θα πρέπει να σεβαστούμε το πλαίσιο του ΠΟΕ και τη μόδα που υπάρχει στον ΠΟΕ. Αλλά το ερώτημα μου παραμένει. Έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα. Θεωρείτε ότι πρέπει κάποια στιγμή ενδεχομένω μπορεί να πρέπει να κλείσουν οι αγορέ μα απέναντι στι αυτές. αυτέ να επαναλάβω κάποια τα σχόλια των συναδέλφων για το γεγονός ότι χαιρόμαστε που η διαδικασία είναι ανοιχτή και διαφανής. Ε, για την, συγγνώμη για τη φωνή μου, η οποία είναι βραχνή. Ε, είναι μετά από την γρήπη του TTIP. Δύο ερωτήσεις. Πρώτον, η, η μέρα εμπορικής πολιτικής. Ενδιαφέρουσα μέρα, μου φάνηκε. Μια ανοιχτή διαδικασία Καλό είναι για να αναπτύξουμε αυτή την πολιτική, να την εξηγήσουμε. Ο, ο Καρλ Μπράουνερ, ο αναπληρωτή Γενικό διευθυντής ε, τη Γενική Διεύθυνσης Εμπορίου, είπε ξεκάθαρα σε ένα πάνελ που συμμετείχα ότι ο πελαπλασιασμός των διμερών συμφωνιών ανά τον κόσμο δεν προωθούν τι πολυμερει ε, συμφωνίε, αλλά παρεμποδίζουν τι πολυμερει συμφωνίε και υποσκάπτουν τι διαπραγματεύσει των ΠΟΕ. Ποια είναι η άποψή σα για αυτή την ε, διατύπωση και πώ θα εξασφαλίσουμε ότι κρατάμε ψηλά τον πολυμερισμό, τις πολυμερίες διαπραγματεύσεις και συμφωνίες. Επίσης, μου άρεσε ότι οι ευρωπαϊκές αξίες και η βιώσιμη ανάπτυξη είναι ψηλά στην ατζέντα σας. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξουμε την προπτική μας από ένα μοντέλο πίεση των ομοτήμων, ας πούμε, ε, και να πάμε σε αναζήτηση άλλων τρόπων. Να μην κάνουμε απλώς ε, ωραία λόγια, δηλώσεις κτλ. Να προ προωθήσουμε πολιτικές συγκεκριμένες που βελτιώνουν πραγματικά τη ζωή των απλών ανθρώπων στον κόσμο ολόκληρο. Ευχαριστώ. Η Έμα. Ευχαριστώ, Επίτροπε, για τα σχόλιά σας. Χαίρομαι που οι αξίες είναι στο επίκεντρο της ομιλίας σας. Και μιλάτε για ανοιχτέ αγορές και ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί απέναντι σε όλο τον κόσμο παρά τα σχόλια που άκουσα από του συναδελφού μα, εγώ πιστεύω ότι δεν μπορούμε να ζούμε εν κενό. Η αποδοσμιοποίηση είναι πραγματικότητα και πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό. Έχουμε τη δυνατότητα μάλιστα να είμαστε ηγέτε, να παίξουμε ηγετικό ρόλο σε όλη αυτή τη διαδικασία. Ελπίζω ότι θα αναπτύξουμε τρόπου για να απλωστευτεί το εμπορικό περιβάλλον και ότι θα βασιζόμαστε σε κανόνε ελευθέρου εμπορίου και όχι κανόνε που του επιβάλλουμε από πάνω προ τα κάτω. Ελπίζω να δούμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Θέλουμε χρονοδιαγράμματα, προθεσμίες. Καθόμαστε στο, καθίσαμε στο τραπέζι και τώρα θέλω να ολοκληρώσουμε αυτές τις συμφωνίες, θέλω να προχωρήσουμε από τις ελπίδες και τα ευχολόγια στο θα κάνω και κάνω. Και πιστεύω ότι έτσι μπορούμε να αλλάξουμε την κατεύθυνση του, της επικοινωνίας μας, της, ε, τη φρασιολογία που χρησιμοποιούμε πρέπει να είναι πολύ πιο ε, έτσι, στεναρή, να έχουμε εμπιστοσύνη Χαίρο, χαίρομαι που αναφέρατε επίσης και την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Θέλω να υπάρξει άνοιγμα προς το Μεξικό και τη Χιλή και να κοιτάξουμε και άλλες περιοχές του πλανήτη. Ελπίζω ότι έχετε τους πόρους που χρειάζεται για να προωθήσετε τη στρατηγική που μας παρουσιάσετε. Θα ήθελα να ακούσω περισσότερα για τη συνολική στρατηγική σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη και τη θέση απασχόληση, πώ θα τα καταφέρει και να αντιμετωπίσουμε και τα άλλα προβλήματα που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μέσω του εμπορίου φτώχεια, παραδείγματο χάρη, και μείωση τη φτώχεια. Αυτά τα δύο, εμπόριο και μείωση τη φτώχεια, πάνε μαζί. Αν θέλουμε ε, αν πολλαπλασιασμό των θέσεων απασχόληση, πρέπει να μειώσουμε τη φτώχεια παγκόσμια. Έχουμε ευθύνη να ανοίξουμε το εμπόριο και να το κάνουμε ελεύθερο εμπόριο. Το θέμα είναι να μπορούμε και να το κάνουμε. Ο κύριος Μπούχνερ παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ Επίτροπε που ήρθατε στην Επιτροπή μας και έχουμε αυτή τη συζήτηση. Επιτρέψτε μου να συνεχίσω σε αυτά τα οποία είπε προλαλήσασα. Είπατε, λέτε, ότι το εμπόριο αυξάνει την παραγωγικότητα. Σίγουρα αληθεύει αυτό. Όμως η παραγωγικότητα και η αύξησή της δεν σημαίνει αυτόματα περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Το αντίθετο η θεωρία στην νεοφιλελεύθερη οικονομία προϋποθέτει διάφορους όρους και προϋποθέσεις για να υπάρχει πλήρης απασχόληση και αυτοί δεν υλοποιούνται. Παράδειγμα, Μεξικό όπου εκατομμύρια, δύο εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης απολέστηκαν. Πώς θα διασφαλίσετε λοιπόν να μην συμβεί κάτι τέτοιο στην Ευρώπη. Δεύτερο, είπατε πιο πριν ότι η νέα εμπορική σας πολιτική τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου θα τα προαγάγει. Μέχρι σήμερα ουσιαστικά δεν τα καταφέραμε. Ας πάρουμε ένα παράδειγμα μεταξύ πολλών, τη Δυτική Σαχάρα. Δεν τα καταφέραμε με βάση τις εμπορικές σχέσεις να καταφέρουμε κάτι. Για τη δημοκρατία μπορώ να πω αυτή η ειδική μορφή που τονίζουμε της ρυθμισμένης συνεργασίας όπως από πλευράς TTIP στοχεύουμε να γίνει είναι ουσιαστικά μια πολύ σημαντική απώλεια δημοκρατίας. Πώς θα αντιμετωπίσετε αυτά τα προβλήματα λοιπόν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Φυσάς παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, δύο θέματα. Ε, μας ικανοποιεί ότι θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις μας με την, την Ισία. Θα ήθελα να εμβαθύνουμε περισσότερο σε αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι την Ισία είναι μία από τις λίγες χώρες, αραβικές χώρες στη Μεσόγειο, που μπορούν με αυθεντική δημοκρατία που έχουν να προχωρήσουν ένα είδος πρόγραμμα Marshall πρέπει να έχουμε για μια μικρή χώρα σαν την Τινησία. Δεν πρέπει να την εγκαταλείψουμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία περνάει αυτή τη στιγμή. Κάποια σημαντική προσπάθεια πρέπει να κάνουμε. Να υποστηρίξουμε λοιπόν την Τινησία που επιπλέον είναι υπόδειγμα, παράδειγμα για πολλές άλλες χώρες. Δεύτερο σημείο που θα ήθελα να σχολιάσω. Με ικανοποίησε πολύ το ότι έγινε λόγος απόψε για τα δικαιώματα του ανθρώπου που εισαχθούν Στι ε, διάφορες ε, ρήτρε συμφωνιών εμπορίου. Ερώτησή μου, πώς μπορούμε να ανταγωνιστούμε με χώρες που δεν σέβονται αυτά τα δικαιώματα, όπως την Κίνα. Για παράδειγμα, σε σχέση με την Αφρική, πολλέ φορές ακούω τα σχόλια ότι εμείς ε, ζητούμε και έχουμε απαιτήσει που άλλες χώρες όπως η Κίνα δεν σέβονται αυτές τις απαιτήσεις για τα δικαιώματα του ανθρώπου. Κάνουν ένα dumping περιβαλλοντικό και κοινωνικό dumping οι Κινέζοι και δεν θα είναι εύκολο να ανταγωνιστούμε με αυτούς υπό αυτούς όρους και προϋποθέσεις. Ποια στρατηγική πρέπει να ακολουθήσουμε σε σχέση με την Κίνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επιτροπέ για τις εξηγήσεις που μας δώσατε. Τέσσερις ερωτήσεις. Πρώτον, έχουμε την τύχη όταν είμαστε βουλευτέ, να δουλεύουμε σε διάφορε κοινοβουλευτικέ επιτροπέ Και εγώ είμαι στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση, α πούμε. Το εμπόριο όντω μπορεί να είναι θετικό για να προωθήσει την ανάπτυξη και δεν το αμφισβητούμε. Δημιουργεί ανάγκε, ανάγκε προσαρμογή, προετοιμασία, κανόνων, ρυθμίσεων. Το ερώτημα που θέτω είναι, είμαστε έτοιμοι ως Ευρωπαίοι να αντιμετωπίσουμε όλες τις εμπορικές συμφωνίες, κάθε είδους. Οι βιομηχανικέ πολιτικές μας ε, οι πολιτικές της εσωτερικής αγοράς είναι έτοιμες, οι κοινωνικές μας πολιτικές είναι έτοιμες, υπάρχουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για την ευρωπαϊκή ανάπτυξη μόνο μέσω του εμπορίου. Πρέπει να κάνουμε επενδύσεις και σε άλλους πυλώνες ανάπτυξης. Ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να συζητήσουμε με τους επιτρόπους που ασχολούνται με αυτές τις άλλες πολιτικές και να δούμε πώς το εμπόριο και οι υπόλοιπε πολιτικές μπορούν να αλληλεπιδράσουν ούτω ώστε να είμαστε πιο δυνατοί και να υπάρξει μεγαλύτερη ευρωπαϊκή ανάπτυξη. Δεύτερο ερώτημα. Για τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένε χώρες. Δεν βλέπω να είναι συνεκτική η πολιτική σας. Η πολιτική ανάπτυξης και η εμπορική πολιτική κανονικά πρέπει να πηγαίνουν χέρι-χέρι. Στα πλαίσια των ε, ε, διαγωνισμών, ας πούμε, ή μάλλον τη αναπτυξιακής πολιτικής, συγγνώμη, συχνά ε, κάνουμε λάθη. Η εμπορική πολιτική δεν υποστηρίζει την απτυξιακή πολιτική. Επίσης, μιλήσαμε πολύ ε, για την εμπορική πολιτική στα πλαίσια τη επίλυση διαφορών. Καταρχά, θα ήθελα να σα μιλήσω για την ε, συμφωνία συνεργασία με το Ισραήλ. Στο κείμενό σα δεν μίλησατε καθόλου γι' αυτό. Νομίζω το εμπόριο θα πρέπει να μα βοηθήσει στην ανάπτυξη, την αμοιβαία ανάπτυξη. Αλλά θα πρέπει επίση να είναι και ένα εργαλείο το οποίο μα επιτρέπει να εξασφαλίσουμε ειρηνιστικές διαδικασίε. Η Συμφωνία συνεργασία με το Ισραήλ μπορείτε να πείτε ότι βελτιώνει την ε, διαδικασία ειρήνη στην περιοχή. Τέταρτο ερώτημα. Οι Ευρωπαϊκέ Αξίε που υποτίθεται ότι προασπίζεστε. Ω ε, Ευρωπαίοι δεν θα, πρέπει, θα πρέπει να δεχτούμε στην, ε, στον ευρωπαϊκό χώρο όλα τα προϊόντα ε, τις που είναι κατάλληλα για κατανάλωση και όταν μιλάω για ακατάλληλη κατανόηση δεν είναι μόνο για την υγεία των Ευρωπαίων, αλλά και την υγεία των άλλων, έτσι, των υπόλοιπων μη Ευρωπαίων. Τι γίνεται με την υποχρεωτική χνηλασιμότητα που μας επιτρέπει ε, να μην προωθούμε ε, τις συγκρούσεις, να μην τροφοδοτούμε τις συγκρούσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επίτροπε, ευχαριστώ για τις πληροφορίες σας. Και ευχαριστώ και για τον ε, σεβάθος διάλογο που έχετε με την Κοινοβουλευτική μας Επιτροπή. Δεν είναι δυνατόν σε ένα λεπτό, σε μια τέτοια παρέμβαση τόσο σύντομη να εμείνει κανεί σε όλα τα θέματα. Το νέο παγκόσμιο εμπόριο αφορά και τι διαπραγματεύσει, αλλά πρέπει να διαπραγματευόμαστε με του εταίρου μα αλλά και να έχουμε διάλογο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω έχετε δίκιο στο ότι η νέα στρατηγική για το εμπόριο πρέπει να προσφέρει αυτά τα εργαλεία για την προαγωγή των αξιών μας υπό πλαίσιο διαφάνειας, υπό ένα ανοιχτό πλαίσιο με συγχωρείτε που ε, λέω αυτά τα γνωστά θέματα, αλλά πρέπει και σε ένα πλαίσιο ε, συζήτησης για τα συμφέροντα της ευρωπαϊκής οικονομίας και τα συμφέροντα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να διεξαγάγουμε, ώστε να προαχθούν αυτά και να προστατευτούν. Και υποστηρίζουμε την πρόθεσή σας να υπάρξει απλούστευση ε, των διαδικασιών, αλλά επίσης και στις διμερείς συμφωνίες εμπορίου που πρέπει να προχωρήσουμε και να δούμε τι θα γίνει με τις διμερείς συμφωνίες εμπορίου μεταξύ των κρατών που είναι κράτη-μέλη, για παράδειγμα στην Ανατολική, και στην έναν της Ανατολικής Ευρώπης και για τις προσδοκίες των μελών της Επιτροπής όσον αφορά την Ταϊβάν και να δούμε τι θα γίνει με τις διαπραγματεύσεις σε σχέση με την Ταϊβάν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε για την παρέμβασή σας και για το ότι παρακολουθείτε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι το μέλλον της ευρωπαϊκής εμπορικής πολιτικής θα εξαρτηθεί από το αν θα είμαστε ικανοί όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα να επεξηγήσουμε στους πολίτες μας ότι αυτό που κάνουμε θα βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσής τους και το, την ποιότητα ζωής τους μέσα στα ίδια τα σύνορά μας σε σχέση με τους εταίρους μας και γι' αυτό είναι σημαντική αυτή η στρατηγική να διαφοροποιήσουμε ποιε πολιτικές και με ποιο τρόπο θα τις ακολουθήσουμε συμμερίζομαι για τη σπουδαιότητα που έχει η διαφάνεια, αλλά πρέπει να έχουμε και τις μελέτες, μελέτες επιπτώσεων εξ άντε και εξ post, για να ξέρουμε ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των εμπορικών πολιτικών και τα αποτελέσματά τους, για να εμβαθύνουμε σε αυτά και να δούμε ότι επίσης συνεπάγεται τη συμμετοχή εκείνων αυτές οι πολιτικές που θα επωφεληθούν από αυτές τις διαδικασίες. Μας αφορά άμεσα και το θέμα της TTIP και πρέπει να μάθουμε από τα σφάλματά μας για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Όσον αφορά για την πολιτική αυτή, η πολιτική εμπορίου, διεθνούς εμπορίου, συμμερίζομαι την άποψή σας για το μέσο ε, που πρέπει να δημιουργηθεί την απασχόληση και την απασχόληση ποιότητας. Αλλά πρέπει να υπάρχει και η παρακολούθηση με άλλες πολιτικές για την προαγωγή αυτού του ε, στόχου. Τεχνολογική πολιτική για παράδειγμα. Δεν θα ωφελούσε να μην έχουμε προσκόμματα στην πολιτική μας αν δεν θα ήταν ανταγωνιστικές οι επιχειρήσεις μας στην παγκόσμια αγορά. Και είναι θεμελιώδες να έχουμε μια πολιτική που θα ενισχύει τα εργασιακά θέματα, τις εργασιακές ψηφιακές προδιαγραφές και να δώσουμε συνέχεια σε αυτή την προσπάθεια. Ως προς αυτά θα ήθελα να μου πείτε πώς θα συντονίσετε αυτά με άλλες πολιτικές και πώς θα μπορέσουμε τα κεφάλαια αυτά να προαχθούν. Ευχαριστώ. Thank you. I'm really not sure what European... Δεν είμαι σίγουρη τι εννοούμε όταν μιλάμε για εμπορική πολιτική, αλλά θα ήθελα να κάνω ένα επικοδομητικό ερώτημα για την πολυπλευρικότητα. Τι συγκεκριμένα μέτρα προβλέπετε ώστε να προωθήσετε την πολυπλευρικότητα φαντάζομαι ότι με όλες τις διμερείς συμφωνίες που υπάρχουν χάνουμε και μια άλλη έννοια που ίσχυε πριν την εμπιστοσύνη τι θα κάνετε λοιπόν συγκεκριμένα για να υποστηρίξετε την πολυπλευρικότητα της Ένωσης. Τέλος ο κύριος Μάτου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ Επίτροπε. Μια σύντομη αναφορά για τις υπερπεριφερειακές περιοχές της Ισπανίας, Γαλλίας και Πορτογαλίας ε, όπου γνωρίζουμε ότι υφίσταται το θέμα στη συνθήκη και επανειλημμένα έχουμε αναφέρει ότι πρέπει να υπάρχουν μελέτες επιπτώσεων για τις επιπτώσεις που θα έχουν οι συμφωνίες αυτές ακριβώς σε αυτές τις υπερπεριφερειακές περιοχές πολύ απομακρυσμένες από την Ευρώπη. Πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον με αυτές τις περιφέρειες και ιδιαίτερα αν συμπεραίνουν ότι θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις σε αυτές οι μελέτες θα πρέπει αντισταθμιστικά μέτρα να υιοθετηθούν ώστε να βελτιωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επίτροπε, μπορείτε να απαντήσετε τώρα. Είστε εδώ σήμερα, πριν ολοκληρωθεί η έκθεση και πριν περάσει, ολοκληρωθεί η διαδικασία, είναι για να ενσωματώσω τις απαντήσεις σας. Δεν έχουμε όλες τις απαντήσεις σήμερα, αλλά ο σκοπός της ανακοίνωσης είναι να μας δείξει πώς το εμπόριο μπορεί να βελτιώσει τη ζωή των Ευρωπαίων, αλλά και των υπόλοιπων λαών, να βελτιώσει την οικονομία, να βελτιώσει και να αναπτύξει επενδύσεις και τι θέσει απασχόληση, αλλά και να λειτουργήσει ως εργαλείο για να προωθήσει αξίες και πολιτικές. Και για να γίνει αυτό με πιο συνεπή και στρατηγικό τρόπο, εμείς ως Κομισιόν δουλεύουμε σε οργανώσεις, σε ομάδες, ούτω ώστε η αναπτυξιακή πολιτική, η εξωτερική πολιτική, η εμπορική πολιτική να είναι πολύ πιο συναφής Συνεπεί μεταξύ τους και να ξεπεράσουμε τα, εμπόρια, τα εμπόδια όσο μπορούμε. Φυσικά το εμπόριο δεν μπορεί να δημιουργήσει ειρήνη στη Μέση Ανατολή ή να εξασφαλίσει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα γίνονται σεβαστά παντού στον κόσμο, αλλά μπορεί να παίξει το ρόλο του. Και μπορούμε να ενισχύσουμε το ρόλο του εμπορίου προ αυτή την κατεύθυνση. Για το πολυμερές επίπεδο, ο κ. Γκασπάρη και άλλοι μίλησαν γι' αυτό. Σύμφωνο ότι το πολυμερές επίπεδο διαπραγμάτευση είναι πολύ σημαντικό. Η κυρία Κέλλερ μίλησε επίσης γι' αυτό και πολλοί άλλοι. Τι προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. πρόθεσμα είναι να δώσουμε την ευρωπαϊκή υποστήριξη για, ε, για να ολοκληρωθεί ο γύρος της Δόχα, ούτως ώστε να μην το χρεωθούμε εμείς, να μην είναι εξαιτία της Ευρώπης. Ε, συνεργαζόμαστε με τη γραμματεία, ε, με συνεργάτες από τον κόσμο, ούτως ώστε να φτάσουμε σε μια ατζέντα που θα συμφωνήσουμε. Μια ατζέντα που θα αφορά την απλούστευση και διαφορετικό επίπεδο φιλοδοξίας ε, από αυτό που απέτυχε πριν από 15 χρόνια. Είναι τελευταία ευκαιρία. Εάν τα καταφέρουμε στο Ναϊρόμπι, ο γύρος της Ντόχα θα πεθάνει. Και αυτό θα είναι πολύ επώδυνο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Και τι, τι άλλο κάνουμε σε πολυμέρες επίπεδο οι πολυμερές συμφωνίες προσπαθούν να ενταχθούν στον ΠΟΕ, ε, ενθαρρύνοντας τα μέλη των ε, συμφωνιών ΤΙΖΑ και τα λοιπά να ενταχθούν, ούτως ώστε να έχουμε μια κρίσιμη μάζα για να μπει αυτή. Ε, συνεργαζόμαστε με τον κύριο Αζερβέντο και με άλλους συνεργάτες για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε συμφωνίες μετά την Τόχα, με ή χωρίς την Τόχα. Χρησιμοποιούμε δηλαδή τον ΠΟΕ ως εργαλείο. Γιατί ο ΠΟΕ δεν μπόρεσε να πετύχει σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό έχουμε όλε αυτέ τι διμερείς συμφωνίε οι οποίε πολλαπλασιάζονται όλο και περισσότερο. Για τότε τι είπα, κύριε Γκασπάρη. Οι Αμερικανοί παρακολουθούν ε, τη δουλειά που κάνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, παρουσια, ε, παρακολουθούν τι ψηφοφορίε, νομίζω ότι μελέτησαν τα ψηφίσματά σα, ε, με κάθε λεπτομέρεια, όλη, κάθε κεραία τη γνωρίζουν. Ε, η διαπραγμάτευση ξεκινάει σήμερα και ίσως μιλήσουν ε, και για αυτά. Αλλά σίγουρα μετά το καλοκαίρι όταν συναντηθούμε με τον ε, πρέσβη Φρόμαν θα μπει το θέμα αυτό επιτάπητος για τη ΣΥΤΑ. θα, ολοκληρώσουμε τα νομικά θέματα, θα περάσουμε στην ε, μετάφραση ε, το καλοκαίρι, ούτω ώστε να μπει στο τραπέζι του Συμβουλίου μετά το, το καλοκαίρι και σε, αρχέ, και σε εσά, το δικό σας τραπέζι, αρχές του επόμενου χρόνου. Ε, πολλοί από εσά μίλησατε για την Κίνα προχωρούμε προς μια επενδυτική συμφωνία. Υπάρχει πρόοδος, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει. Ε, με το Βιετνάμ. Είμαστε κοντά στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία οριστικοποίηση, αλλά είμαστε πολύ κοντά με την Ιαπωνία. Προχωράμε. Είχαμε μια συνοκορυφή με την Ιαπωνία πριν από κανένα μήνα στο Τόκιο και συμφωνήσαμε με τους διάφορους υπουργού και τον Πρωθυπουργό να ολοκληρώσουμε τις, να επιταχύνουμε τις συζητήσεις και να κάνουμε όσο περισσότερα βήματα μπορούμε πριν το τέλος του 2015. Ταϊβάν. Είναι ένα θέμα το οποίο εξετάζουμε. Και θα μιλάει και γι' αυτό η ανακοίνωση. Και ξέρω ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται πάρα πολύ, τουλάχιστον κάποιοι ευρωβουλευτέ για αυτό το θέμα. Και αν θα μπορούσαμε οι σχέσει με την Ταϊβάν να πάνε παραπέρα. Για τους θελωνιακούς κανόνες. Ε, είναι Ευρωπαϊκή αρμοδιότητα, αλλά την εφαρμογή την έχουν τα κράτη-μέλη. Είναι ευθύνη των κρατών μελών. Εδώ συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη ε, με βάση τι βέλτιστε πρακτικέ. Είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να εφαρμόσουν την εμπορική πολιτική τα κράτη-μέλη και πρέπει να εστιάσουμε στο πώ θα γίνει αυτό πολύ πιο συνεπέ ε, μέσω τη ανακοίνωση. Να ενισχύσουμε βεβαίω την τελωνιακή συνεργασία, ε, η οποία τελωνιακή συνεργασία θα ε, διευκολύνει το εμπόριο. Και η συμφωνία του Μπαλί για τη διευκόλυνση του εμπορίου είναι καλό παράδειγμα για το πώ μπορούμε να συνεργαστούμε σε πολυμερέ επίπεδο. Κυρία Μόσκα, μιλήσατε για το θέμα της ε, προσπελασιμότητας, της διαφάνειας. Ο στόχος είναι αυτή η στρατηγική να είναι ευρεία. Και να μην το διαβάσουμε μόνο εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα του εμπορίου. Τέλο πάντων, παρότι δεν είναι και best seller, τουλάχιστον ο κόσμο να μπορεί να διαβάσει αυτό το κείμενο, αυτή τη συμφωνία και να μάθει για τη δουλειά που γίνεται για τα εμπορικά θέματα και την εμπορική πολιτική. Είναι σημαντικό να έρθουμε σε επαφή με τον κόσμο, να υπάρχει διαφάνεια, να, εξη, εξηγήσουμε το ρόλο του εμπορίου στην οικονομία, στην παγκοσμιοποίηση, προ όφελο των καταναλωτών. Για τα πράσινα αγαθά και τι κλιματικέ συζητήσει. Τα, τα πράσινα αγαθά μπορούν να βοηθήσουν εκεί. Μπορούμε να Ελπίζω να πετύχουμε μια πρώτη συμφωνία επί ενό καταλόγου που θα είναι έτοιμο το Δεκέμβριο, ούτω ώστε να μπει στη διαδικασία του Παρισιού. Αγαθά λοιπόν τα οποία θα εξαιρεθούν από τα τελωνία και υπηρεσίε που θα μας βοηθήσουν τόσο ώστε να πετύχουμε τους στόχους ε, καταπολέμησης κλιματικής αλλαγής και βιώσιμης ανάπτυξης. Κάμπολ, για την Ινδία. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, είχαμε μια συνάντηση με τον Υπουργό στο Παρίσι πριν από κάνα μήνα. Συμφωνώ ότι ναι, όντω θα συναντηθούν οι βασικοί διαπραγματευτέ τον Αύγουστο για να δούμε πού βρισκόμαστε, για να δούμε αν υπάρχουν τρόποι για να προχωρήσουμε. Ξέρουμε ότι έχουμε δυσκολίε με την χώρα αυτή, αλλά ελπίζω τουλάχιστον να έχουμε μια επικοδομητική συνάντηση και να δούμε πού θα μα οδηγήσει. Ελπίζω να επανέλθω με περισσότερε πληροφορίε σε εσά που είστε εισηγητή, αλλά και στην Επιτροπή σα γενικά, για να σα πω ποιο είναι το αποτέλεσμα των συναντήσεων αυτών. Αυστραλία-Νέα Ζηλανδία. Πολλέ επαφέ είχα με του εκπροσώπου των χωρών αυτών για να δούμε πού βρισκόμαστε. Φυσικά έχει πολιτική σημασία να εμβαθύνουμε τις σχέσεις με τις χώρες αυτές. Αλλά πριν προχωρήσουμε σε διαπραγματεύσεις για συμφωνίες, να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε το ίδιο επίπεδο φιλοδοξίας. Και εμείς και εκείνοι. Και αυτή η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και ελπίζω να μπορέσουμε να κάνουμε μια πρόταση, κατά πάσα πιθανότητα, τον Οκτώβριο μέσα της ανακοίνωσής μας. Κυρία Σάκε, πώς μπορούμε να προωθήσουμε τι αξίες μας. Ε, αυτό είναι ολόκληρο σεμινάριο. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε σε ένα σεμινάριο. Ο στόχο τη ανακοίνωση είναι να κάνουμε μια στρατηγική προσπάθεια σε αυτό το επίπεδο. Όπω ε, βεβαίως το εμπόριο, όπω είπαν ε, η κυρία Μακλάρκιν και άλλοι, είναι οικονομικό εργαλείο. Το θέμα είναι πώ θα συνεργαστούμε, θα εξασφαλίσουμε μια συνεργασία ανάμεσα στην αναπτυξιακή πολιτική, την εξωτερική πολιτική και την εμπορική πολιτική, ούτω ώστε να προωθήσουμε την ανάπτυξη προ μια κατεύθυνση που να συνάδει και να προωθεί τι αξίε μα. Για να το κάνουμε αυτό, θα πρέπει να υπάρχει πιο ηγετικό ρόλο. Το Κοινοβούλιο ε, αποφάσισε να δώσει μεγάλη σημασία στην ε, κοινοβουλευτική αυτή επιτροπή εμπορίου. Ε, δίνεται μεγάλη έμφαση. Βλέπετε πόσο κόσμο έχει αυτή η επιτροπή. Αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να κάνουν το ίδιο. Γιατί η εμπορική πολιτική είναι ψηλά στην ατζέντα στη δημόσια συζήτηση. Εσείς κάνετε τη, τη δουλειά σας και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας ως Επίτροποι, αλλά και τα κράτη-μέλη πρέπει να είναι πολύ πιο παρόντα. Ουκρανία. Ολοκληρώσαμε μια τεχνική συνάντηση με προσώπους Ουκρανίας και Ρωσίας για κάποια συγκεκριμένα θέματα που έχουν εντοπιστεί ως πρόβλημα στην DCFTA, στην Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου. Αναλύσαμε τα συμπεράσματα και θα κάνουμε αρχές Σεπτεμβρίου μία συζήτηση πολιτική με τους δύο υπουργούς, τους δύο της Ουκρανίας και της ε, Ρωσίας εμπορίου. Κύριε Σόλτς, μιλήσατε για το εξή. Για το αν δέχονται, το δέχονται τα μέλη. Είχαμε μία συνάντηση σε επίπεδο Συμβουλίου και τα συζητήσαμε με τα κράτη-μέλη. Τα κράτη-μέλη είχαν τη δυνατότητα να πούν, να πούν τις απόψεις τους. Οι συνεργάτες μου και εγώ ακούσαμε και ήρθαμε σε επαφή με πολλά ακούσαμε τις απόψεις τους και νομίζω ότι θα ληφθούν αυτά στην τελική ανακοίνωση. Για τις γεωγραφικές περιοχές, δεν μπορώ να πω σε κάθε χώρα, γιατί τα πράγματα αλλάζουν και θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε. Γι' αυτό μόνο λίγες χώρες θα αναφέρουμε, αλλά είναι θέμα να δούμε τον πλανήτη αναπεριοχές και επίσης και το θέμα των πόρων και από πού προέρχονται. Κύριε Ζαντό, καταλαβαίνω την κατάθλιψή σας. Πολλά από αυτά που είπατε υπονοούσαν την Ελλάδα βέβαια. Αυτό υπάρχει πίσω από τις συζητήσεις μας σήμερα. Αν ακούσατε καλά όμως τι είπα, μίλησα για τις αξίες, για τη δημοκρατία, για τη σημασία του να υπάρχει μεγαλύτερη συνέπεια στην εμπορική μας πολιτική για να βελτιώσουμε τις συνθήκες ζωής του τρίτου κόσμου. Ελπίζω ότι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε, μπορούμε να συζητήσουμε ε, και πολλές φορές μας έχετε δώσει πολλές ιδέες. Και νομίζω ότι θα δείτε ότι θα απεικονιστούν στην ανακοίνωση που θα εκδώσουμε. Κυρία Μπεγκίν. Άκουσα, και απάντησε κάποια από τα πολυμερή θέματα. Για τα πράσινα αγαθά τον ΠΟΕ και το Τσίσα. Μετά τον Παλί βέβαια. Αλλά τώρα μετά την επιτυχή διάσκεψη του Ναϊρόμπι νομίζω ότι τα πρότυπα για τους κανόνες προέλευσης που αναφέρατε είναι ακριβώς το είδος θέματος που θα έπρεπε να συζητάει ο ΠΟΕ, να συζητάμε στον ΠΟΕ. Και γι' αυτό μπορούμε να τα επαναφέρουμε και στο, στη συζήτηση του θέματος της πολυπλευρικότητας. Κύριε Ντεράνς, νομίζω ότι οι ανοιχτές αγορές είναι κάτι καλό και για την Ευρώπη και για όλες τις χώρες του κόσμου, αλλά πρέπει να υπάρχει καλή διαχείριση προφανώς. Το θέμα της γεωργίας τώρα και των γαλακτοκομικών καθώς και των αμπελοϊνικών είναι πολύ ανταγωνιστική τομής και θα, δεν υπάρχει λόγος να μην υποφεληθούν από τις εμπορικές συμφωνίες. Όχι μόνο τη TTIP αλλά και τις συμφωνίες με την Ιαπωνία. Αναφέρατε δύο δημοσκοπήσεις στη Γαλλία, υπάρχουν και άλλες όμως που δείχνουν ότι η εμπορική μας πολιτική την χάνει στήριξη. Το αναφέρει είναι πολιτική που προκύπτει από τις συνθήκες και που έχει εντολή από όλες τις χώρες μέλη, επομένως εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι οι ανοιχτές αγορές είναι κάτι καλό για την Ευρώπη, για τον πολίτη, για τον καταναλωτή. Κύριε Βαλέντσα, για το θέμα της Κίνας. Είναι πολύπλοκο πρόβλημα. Το βλέπουμε και εμείς το εξετάζουμε εσωτερικά στην Κομισιόν. Αν αποφασίσουμε να βγάλουμε την Κίνα από τον κατάλογο, αυτό δεν μπορεί να το αποφασίσει από μόνη της η Κομισιόν. Θα κάνει πρόταση πρώτα στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Θα είναι κοινή πρόταση δηλαδή, αλλά πρέπει πρώτα να τα ξανασκεφτούμε εσωτερικά και εσείς θα τα σκεφτείτε, ξέρω εδώ. Κύριε Κέντον νομίζω ότι απάντησα σε μερικά από τα θέματα που αφορούσαν τον ΠΟΕ. Με αυτόν τον τρόπο συντονίζουμε τα θέματα εμπορίου, ανάπτυξης, για να είμαστε σίγουροι ότι και με τις αναπτυσσόμενες χώρες θα βρισκόμαστε σε ίδιο μήκος κύματος. Θα έπρεπε περισσότεροι επίτροποι να το κάνουν αυτό, εξαιρετική είναι η πρόταση που κάνατε, αλλά προσπαθούμε να επιτύχουμε συνέπεια και συνοχή. Ας πούμε για την Τινησία αυτή την εβδομάδα πολλοί επίτροποι θα συζητήσουν για να στηρίξουμε την εμπορική πολιτική της Τινησίας, τις φοιτητικές ανταλλαγές, τέτοια πράγματα. Έτσι το προσπαθούμε. Δεν λέω ότι το πετυχαίνουμε 100% αλλά προσπαθούμε. Προσπαθούμε. Τώρα για τις ανοιχτές αγορές νομίζω το είπα κυρία Κλάρκιν. Δεν μπορώ να σας δώσω διορίες και χρονοδιαγράμματα αλλά τα προωθούμε, τα προωθούμε. Δεν έχει ημερομηνίε η ανακοίνωση βέβαια γιατί θέλουμε καλή συμφωνία μάλλον παρά γρήγορη. Για την Ιαπωνία, για το Βιετνάμ δεν είναι εύκολο να τα κανονίσουμε γρήγορα γρήγορα. Δεν μπορούμε να βάλουμε συγκεκριμένη ημερομηνία αλλά δεν καθυστερούμε παραπάνω από ό,τι θα έπρεπε. Τα αποτελέσματα τώρα για τα ωφέλη του εμπορίου είναι βασικό θέμα. Γι' αυτό μίλησα για τη σημασία της εφαρμογής στενότερης συνεργασίας με τα κράτη-μέλη και με ως εποπτικό σώμα για την όντως εφαρμογή των συμφωνιών και για να υπάρξουν πραγματικά ωφέλη και υπάρχουν και τα παραδοσιακά εργαλεία του εμπορίου όπως οι κανόνες του ΠΟΕ και άλλα εργαλεία με τα οποία να οθήσουμε τους εταίρους μας να έχουν αποτελέσματα. για τι σα είπα, για την Τινησία είπα, για το Ταϊβάν νομίζω είπα επίσης, ε, μετά η κυρία Κέλλερ, τι να κάνουμε συγκεκριμένα για την πολυπλευρικότητα, νομίζω απάντησα και γι' αυτό. Νομίζω τα είπα όλα κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την καταπληκτική συζήτηση με τις τόσο ενδιαφέρουσες ιδέες και αν μου επιτρέπετε πρόεδρε θα ήθελα και εγώ να σας ευχηθώ καλάς διακοπάς που μας αξίζουν όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλους. Και... Για την συνέχεια που θα δώσουμε χρειάζεστε κάποια ξεκούραση και θα ξανασυναντηθούμε μετά τις θερινές διακοπές. Σας ευχαριστούμε πολύ Επίτροπε. Uh, Good. Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt. Πολύ καλά περνάμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης η προσχώρηση του Εκουαδόρ του σημερινού στην Συμφωνία Εμπορίου όπως ε, της Κολομβίας και του Περού. Ιούνιο 2014 ολοκληρώθηκε και <clears throat> μονογράφηκε το Δεκέμβριο 2014 και τώρα πρόκειται ησυχία παρακαλώ για την υλοποίηση αυτής της ε, προσχώρησης και με αυτό θα ασχοληθούμε και ο εισηγητής μας έχει ένα ψήφισμα το οποίο έχει σχεδιάσει, έχει τον λόγο για να μας το παρουσιάσει. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ποια είναι η αφετηρία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα <clears throat> πολυμερές εμπορικό ε, με το Περού και την ε, ε, Κολομβία και η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν αβέβαια για αυτή τη συμφωνία. Έγινε όμως υπό τον όρο ότι συγκεκριμένα βήματα και διαβήματα θα αναλαμβανόντουσαν ώστε η κοινωνική κατάσταση και τα δικαιώματα του ανθρώπου θα προστατευόντουσαν και θα βελτιωνόταν η κατάσταση συνολικά. Η προσχώρηση του η σε αυτή τη συμφωνία δεν αλλάζει αυτούς τους ε, βασικούς στόχους. Το αντίθετο, η προσχώρηση είναι μια σημαντική χρονική στιγμή να εξετάσουμε αν οι όροι αυτοί για αυτή τη συμφωνία πράγματι διαφυλάσσονται και κοινωνικά και οικονομικά. Τα πρώτα αριθμητικά στοιχεία που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη αυτού του εμπορικού πλαισίου με την Κολομβία και το Περού παραμένουν πολύ πίσω από τις προσδοκίες μας. Χαίρομαι ότι η κυβέρνηση του Ισημερινού συμμερίζεται τις απόψεις μας για τα κοινωνικά θέματα και γι' αυτό ρητά θα ήθελα να ευχαριστήσω για την επιστολή του Υπουργού Εμπορίου που νομίζω την έχετε όλοι στα χέρια σας, που αναφέρεται στους στόχους και τα κεκτημένα της κυβέρνησης και τα τονίζει συνειδητοποιούμε από την υλοποίηση της συμφωνίας με την Κολομβία και το Περού και την Κεντρική Αμερική υπάρχει μεγάλη πίεση ανταγωνισμού για τις εξαγωγές προϊόντων του σημερινού και υπάρχει η ε, επιθυμία να υπάρξει ένα ισότιμο πλαίσιο για τον Ισημερινό για αυτά τα προϊόντα. Δεν θα καθυστερήσει το ψήφισμά μας αυτές τις διαργασίες. Όμως με αυτό το ψήφισμα θα υλοποιήσουμε τις ευθύνες μας ως Ευρωκοινοβούλιο για αυτούς τους τομείς και θα καταδειχθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στα κράτη-μέλη που υπάρχουν ανάγκες να δράσουμε ώστε να είναι πιο αποτελεσματική η συμφωνία, ώστε ο πληθυσμός και στις δύο αυτές περιοχές να υποφεληθεί. Γι' αυτό ζητεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το ψήφισμα ταχαίως να υποβληθεί μια ανάλυση για την υλοποίηση και τα επιτέγματα της συμφωνίας. Η κυβέρνηση του σημερινού ζητείται με αυτή την αφορμή την εμπειρία του, της Κολομβίας και του Περού να την αναλύσουν ώστε από κοινού να δούμε οι μέχρι σήμερα κοινωνικές επιτυχίες μπορούν να επηρεάσουν τους όρους αυτής της εμπορικής συμφωνίας και πώς μπορούν να επεκταθούν. Και υπό αυτό το σκηνικό επισημαίνει το ψήφισμα το, τη σύσταση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας. Μια σαφής αξιολόγηση για τον Ισημερινό δίνει επίσης και την επέκταση των εξαγωγών προς την Κολομβία και το Περού, ιδιαίτερα μέσω της Κολομβίας, την ενισχυμένη δηλαδή εμπλοκή των ΙΠΑ σε σχέση με την Κολομβία και την επέκταση των δραστηριοτήτων τους όσον αφορά επιχειρήσεις των ΙΠΑ που δραστηριοποιούνται εκεί. Αυτό έχει και επιπτώσεις ε, για τον πληθυσμό της ε, Υπέθρου, ιδιαίτερα τους μικροαγρότες και κατά των γηγενών πληθυσμών, αλλά επίσης και κατά του περιβάλλοντος. Γι' αυτό ζητεί το ψήφισμα από κοινού με το Εκουαδόρ, με τον Ισημερινό, να μεριμνήσουμε για αυτά τα θέματα. Θα χαιρόμουν αν η κυβέρνηση του Ισημερινού με τη μεγάλη πραγματογνωμοσύνη της και με τις μεγάλες επιτυχίες κατά τα τελευταία 8 χρόνια αν αναφερόταν σε ένα κατάλογο συνοδευτικών μέτρων για αυτή την εμπορική συμφωνία που η υλοποίησή τους με την υποστήριξη της Ευρώπης θα μπορούσε να διασφαλιστεί. Και ταυτόχρονα στην κοινή συζήτηση σε όλες τις χώρες της κοινότητας των Άνδεων να στραφεί η προσοχή σε αυτά τα θέματα όπως το αξίζουν για να αναλυθούν. Γνωρίζουμε ότι δεν εμπλέκονται εξίσου όλοι στην εμπορική πολιτική για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά μέτρα και ότι πολλές φορές υπάρχουν πολλά προσκόμματα εμπορικά. Γι' αυτό θέλουμε για να διασφαλίσουμε τις επιτυχίες και γι' αυτό υποστηρίζουμε την πρωτοβουλία του σημερινού στο πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών με μια σύμβαση να εξεταστεί η δράση των διεθνικών εταιριών ώστε να υπάρξει ένα βελτιωμένο πλαίσιο για αυτές τις δράσεις. Και στρεφόμενοι στο ψήφισμα για την Λατινική Αμερική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την τελευταία κοινοβουλευτική θητεία αναφερόμαστε και πάλι στο μεγάλο ενθουσιασμό που μας ενέπνεε ώστε να μπορέσουμε από πλευρά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να εξετάσουμε το εγχείρημα Γιασούνη, του Εθνικού Δρυμού Γιασούνη. Και από τον Ισημερινό, την Κολομβία και το Περού να προβληματιστούμε και να δούμε πώς τέτοιες προοπτικές ως ιδέες μπορούν πραγματικά να εφαρμοστούν στην κοινωνική ζωή και προς όφελος των πολιτών και του περιβάλλοντος. Λαμβάνοντας υπόψη την διάσκεψη κορυφής των Ηνωμένων Εθνών του Σεπτεμβρίου, μπορεί ακριβώς να δημιουργηθεί και ένα συγκεκριμένος χρονορίζοντας για όλα αυτά. Και έτσι υπό αυτό το πρίσμα τέτοιες πτυχές θα ληφθούν υπόψη για τη μελλοντική εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ψήφισμα θέλει να καταστήσει σαφές ότι στην Ευρώπη και στην κοινότητα των άνδρων πολλά πρέπει ακόμα να γίνουν ώστε οι προοπτικές των ε, πληθυσμών να βελτιωθούν. Το ψήφισμα υπογραμμίζει ακόμα και τη βούλησή μας να πράξουμε περισσότερα προς αυτήν την κατεύθυνση. Θέλω ρητά με αυτή την ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εμπορίου και την κυβέρνηση του σημερινού και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τις πολλές επαφές και συζητήσεις που έδωσαν ευκαιρία να εμβαθύνουμε σε όλα αυτά τα θέματα και να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο με την προσχώρηση του Εκουαδόρ σε αυτή τη συμφωνία να συνδυαστούμε ώστε οι εκπρόσωποι της οικονομίας και τον ΜΚΟ σε σχέση με τον Ισημερινό να δράσουν και θέλω επίσης και να ευχαριστήσω και τους κοιόδης εισηγητές ιδιαίτερα τον συνεισηγητή συνάδελφο Φίσας για την Κολομβία και, τον, ε, και το Περού. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που συμμετείχαν και θα δούμε ποια συνέχεια θα δώσουμε μετά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε ο Φίσας παρακαλώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Πρόεδρε. Ο κύριος Σόλτ είπε ότι πέρυσι τον Ιούλιο ολοκληρώθηκαν διαπραγματεύσεις της εμπορικής συμφωνίας μεταξύ του Εκουαδόρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης με επιτυχία. Διαπραγματεύσεις ε, όπου το Εκουαδόρ εγκατέλειψε το 2009. Και είναι καλά νέα το ότι θα ενσωματωθεί τελικά σε αυτή τη συμφωνία. Νομίζω ότι είναι πραγματικά καλό νέο αυτό. Και για τις δύο πλευρές. Εδώ τώρα συζητάμε την ε, πρόταση ψηφίσματο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την πρόσβαση του Εκουαδόρ στη συμφωνία. Μαζί με τον ε, κανονισμό που θα ολοκληρώσει τη διαδικασία ε, προσχώρησης του Εκουαδόρ. Ευχαριστώ τον κύριο για τη δουλειά που έκανε για σε αυτή την πρόταση ψηφίσματος. Ήθελα να κάνω όμως κάποια σχόλια επί του κειμένου αυτού. καταρχά. νομίζω ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτό το ψήφισμα αφορά την ενσωμάτωση, την ένταξη του Εκουαδόρ στην εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, Κολομβίας και Περού. Και δεν πρόκειται εδώ για μια εξέταση του πώ λειτουργεί η ισχύουσα συμφωνία με την Κολομβία και το Περού. Γιατί γι' αυτό υπάρχει ομάδα παρακολούθηση. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στο ψήφισμα, τα οποία από το 11 έως το 22 νομίζω, όπου γίνεται μια ανάλυση της κατάστασης στο Εκουαδόρ. Πολιτική ανάλυση, ε, περιβαλλοντική ανάλυση. Αλλά όμως δεν είναι ο στόχος αυτού ψηφίσματος, νομίζω, αυτά τα θέματα. Πέρα από τις απόψεις που έχουμε για αυτά τα θέματα, το ψήφισμα νομίζω ότι θα πρέπει να εστιάσει περισσότερο στην αξιολόγηση της ίδιας συμφωνίας. Επίσης, αντίθετα, λείπει μία αξιολόγηση του περιεχομένου του οικονομικού περιεχομένου της συμφωνίας. Ίσως θα πρέπει να, να μπουν τα, τα εμπορικά στοιχεία, τα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη που, πρέπει να έχει, που θα έχει μάλλον η Ευρώπη και το Εκουαδόρ. Μία ερώτηση στον κύριο Σόλτς, γιατί δεν κατάλαβα, εάν προτείνει μια, ένα οδικό χάρτη για το Εκουαδόρ. Ναι ή όχι. Και θα ήθελα να μου το διευκρινίσει παρακαλώ. Επίσης, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία όπου συμφωνούμε και με μικρές αλλαγές θα μπορούσαν να γίνουν απόλυτα αποδεκτά τα σημεία αυτά από την ομάδα μου. Θα ήθελα να σας πω ότι είμαστε στο ίδιο μήκο κύματος με αυτό που υπόθηκε για την μπανάνα, που είναι από τους μεγαλύτερους παραγωγούς μπανάνας και μπορεί οι εξαγωγέ να απειλήσουν τα δικά μας ευρωπαϊκά προϊόντα. Και Χέλμουντ, συμφωνώ ότι πρέπει να σεβαστούμε τις ποσοστώσεις εισαγωγή που αναφέρει η συμφωνία και νομίζω ότι είναι σημαντικό η Επιτροπή να μας ενημερώσει συγκεκριμένα για την εξέλιξη των εισαγωγών μπανάνας και μάλιστα εκ των προτέρων. Και εγώ και ο Χέλμουτ ε, υποστηρίζουμε το σημείο 28. Να διαβάσεις όλες, όλα τις εκθέσεις, όλες τις πράξεις, βέβαια, γιατί είναι μια τεράστια δουλειά. Τέλος πάντων, πρέπει να αρχίσουμε τη δουλειά πάνω σε αυτό το ψήφισμα και να πω ότι εγώ, η ομάδα μας, φυσικά θα υποστρίξουμε απόλυτα την προσχώρηση του Εκουαδόρ στη συμφωνία αυτή. Ευχαριστούμε θέρμα για τους σοσιαλδημοκράτες είμαι εγώ ο συζητητής. Μπορώ να προσθέσω τη φωνή μου στις παρατηρήσεις αυτές. Πράγματι και πολιτικά και οικονομικά η προσχώρηση αυτή είναι κάτι που μπορούμε να χαιρετήσουμε. Και το κάνουμε και αυτό. Και βρίσκω ότι το σχέδιο ψηφίσματος του Helmut Scholz προσφέρει μια σημαντική, σημαντικά στοιχεία για αυτή τη διεργασία και ευθυγραμμίζεται εξάλλου με το ψήφισμα που είχαμε κατά το παρελθόν για την Κολομβία και το Περού και είχαμε προετοιμάσει τότε. Και το θέμα επίσης που στα σημεία 2 και, 2 ε, και 3 και 4 αναφέρονται, τα θέματα δηλαδή της εφαρμογής, της υλοποίησης, πρέπει να τύχουν προσοχής από πλευράς μας. Και σε σχέση με το Περού είδαμε ότι σημαντικές προκλήσεις αντιμετωπίζονται όσον αφορά την εφαρμογή, ιδιαίτερα όσον αφορά την ενημέρωση και πληροφόρηση αυτής της εφαρμογής και υλοποίησης. Και μπορούμε περισσότερα να πράξουμε σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Και το βρίσκω και σωστό ότι στο ψήφισμα η οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη του σημερινού είναι κάτι που τονίζεται. Ιδιαίτερα όσον αφορά την κρίζωση, την μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη του κοινωνικού τομέα, του κοινωνικού κράτους. Και η κυβέρνηση του Εκουαδόρ σημαντικά κονδύλια διέθεσε, νομίζω πάνω από 40 εκατομμύρια αμερικανικά δολάρια, <clears throat> που διέθεσε στον κοινωνικό τομέα. Τώρα, το θέμα της εφαρμογής, της υλοποίησης, της ε, σύμβασης 80 ε, και 98 της ε, Διεθνούς Οργάνωσης, του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας και την ενδυνάμωση των εργασιακών δικαιωμάτων έχει πολύ αποφασιστική σημασία. Και νομίζω αυτό και πάλι σωστά πρέπει εδώ και τονίζεται με τον ε, ενδεδειγμένο τρόπο. Και η μη επικύρωση του 129, δηλαδή της επιθεώρησης και των ελέγχων επιχειρήσεων μέσω εργασιακών ε, ε, επιθεωρήσεων και στο θέμα της Κολομβίας και του Περού αυτό καταδείχθηκε ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση στην Κολομβία και το Περού. Είχαμε έναν οδικό χάρτη δημιουργήσει για αυτά τα θέματα και το θέμα των επιθεωρήσεων εργασίας και εργασιακών θεμάτων και ο αριθμός των επιθεωρητών για αυτές τις επιθεωρήσεις και η συχνότητα των επιθεωρήσεων και ελέγχων όσον αφορά τις επισκέψεις τους σε επιχειρήσεις για δίωξη και κύρωση παραβιάσεων και παραβάσεων είναι μια σημαντική πρόκληση. Και έτσι λοιπόν οι επιθεωρήσεις εργασίας πρέπει ξεχωριστά να αντιμετωπίζονται και να αναφέρονται. Και στην παράγραφο 15 αναφέρεται το θέμα της ευθύνης των επιχειρήσεων και μπορεί κανείς για παράδειγμα να εξετάσει το θέμα του δίκαιου εμπορίου, του θεμητού εμπορίου ξεχωριστά για την Κολομβία ξεκίνησε ένα μικρό πιλωτικό σχέδιο για αυτό το εμπόριο, το δίκαιο εμπόριο, για τα προϊόντα που ε, διοχετεύονται στην αγορά μας, ε, ε, γεωργικά προϊόντα. Θετικό ήταν το εγχείρημα αυτό. Και τέλος, η σκέψη ότι φυσικά θα πρέπει να ενισχύσουμε τις ε, διαδικασίες ώστε να υπάρχει ενισχυμένη διασύνδεση μεταξύ των χωρών της κοινότητας των άνδεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αντιδιαστολή με άλλους που στρέφονται περισσότερο ιδιαίτερα στον χώρο του ειρηνικού και δεσμεύονται ε, και αναπτύσσουν τις προσπάθειές τους σε αυτό το πλαίσιο. Πρέπει να δούμε εκείνα τα κράτη που στρέφονται προς την Ευρώπη από τη Λατινική Αμερική και να τα ενθαρρύνουμε. Αυτές είναι οι πρώτες παρατηρήσεις μου. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Και περνάμε τώρα στη συνέχεια σε εσά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Οι συντηρητικοί δέχονται τις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου, ιδιαίτερα αυτήν εδώ. Την έχουμε υποστηρίξει και το κανονισμό GSP για να καλυφθεί το χάσμα που είδαμε το έλλειμμα μισή χρόνο μέχρι να αρχίσει η πλήρης εφαρμογή αυτής της Συμφωνίας Ελεύθερων Συναλλαγών. Πιστεύουμε ότι αυτό θα βοηθήσει όχι μόνο την ευρωπαϊκή πλευρά για να αυξήσει το εμπόριό της, αλλά και την οικονομία του Ισημερινού για να μειώσει την ανέχεια και να αναπτύξει την οικονομία. Πιστεύουμε λοιπόν πράγματι ότι αυτή η συμφωνία θα μπορούσε να είναι πολύ θετική και για τις δύο πλευρές για την αύξηση επενδύσεων και εμπορίου και επίσης για, ως μοχλός για την οικονομική ανάπτυξη του Εκουαδόρ του σημερινού. Θα ήθελα τώρα να επανέλθω σε αυτά που είπε ο κύριος Φίσας προηγουμένως δηλαδή την ένταξη μιας χώρας σε μια συνθήκη που ήδη προϋπάρχει με την Κολομβία και το Περού. Και αυτό σημαίνει ότι έτσι θα συμπληρωθεί η συμπερίληψη μιας ολόκληρης γεωγραφικής περιφέρειας και δεν θα χρειαστούν χωριστές συμφωνίες. Γι' αυτό δεν πιστεύουμε ότι χρειάζονται πρόσθετες απαιτήσει ούτε πιστεύουμε ότι στη μέση της διαδικασίας έγκρισης πρέπει να αρχίσουμε να ζητάμε δεσμευτικά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη ή να ζητήσουμε από τον Ισημερινό να υποσχεθεί ότι θα σεβαστεί ορισμένους κανόνες για το περιβάλλον ή για τα εργασιακά διότι θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει εταιρικά παρέμβαση σε εσωτερικά άλλης χώρας αν επιβάλλουμε προϋποθέσεις και τους απαιτήσουμε να εφαρμόσουν καινούργιο και χωριστό νομικό πλαίσιο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ακολουθήσουμε εδώ τις παραδόσεις των εταίρων μας και όχι να επιβάλλουμε κάτι. Πάντως, γενικά όπως σας είπα και από την αρχή είμαστε υπέρ και του ψηφίσματος με μορφή που να επιτρέπει την έγκριση της συμφωνίας και όσων έχουν προσυμφωνηθεί. Αυτά έχω να σας πω. Και προσβλέπουμε στις τελικές διαπραγματεύσεις και με τους άλλους κοιόδες Ελπίζω να καταλήξουμε σε βιώσιμους συμβιβασμούς. Ευχαριστούμε πολύ. Από τους φιλελεύθερους ο κύριος Τρεμόσα κανονικά θα ήταν αλλά απουσιάζει. Επομένως η κυρία Κέλλερ. Ευχαριστώ, μπορώ να είμαι σύντομη. Εμείς δεν ήμασταν και τόσο πολύ υπέρ των άλλων συμφωνιών με την Κολομβία και το Περού, αλλά δεν μας ενοχλεί να προσθεθεί και αυτή η χώρα. Απλώς να πάρουμε τα μαθήματα που μας έδωσε η εφαρμογή της συμφωνίας με τις δύο άλλες χώρες. Γι' αυτό θα καταθέσουμε μερικές τροπολογίες. Γενικά όμως συμφωνούμε με τον εισηγητή. Θα καταθέσουμε μερικές τροπολογίες και ελπίζω να υπάρξει συμφωνία και άλλων. Ευχαριστούμε. Τζούντ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να γυρίσω στο θέμα για το κεφάλαιο της αηφόρου ανάπτυξης στον οδικό χάρτη. Εδώ το θέμα της συνεκτικότητας και συνέχεια τίθεται σε σχέση με τρίτες χώρες, σε σχέση μας με τρίτες χώρες και τη θέση του Κοινοβουλίου σε σχέση με τον οδικό χάρτη με την κοινότητα των άνδεων συνολικά. Είναι λοιπόν σημαντικό τα ίδια κριτήρια να ισχύουν για όλες τις χώρες που <clears throat> σε σχέση με τους όρους της συμφωνίας θα πρέπει να συμμορφώνονται και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό διότι είναι σαφές από την Τις τελευταίες αναφορές ε, του ε, Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας ότι υπάρχουν παραβιάσεις όσον αφορά την εργασιακή νομοθεσία σε σχέση με τον Ισημερινό και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίζονται αυτά τα θέματα. Ιδιαίτερα όσον αφορά και το δικαίωμα, το δικαίωμα των εργαζομένων στον κρατικό τομέα να μπορούν να απεργούν. Και είναι κέρια σημασία σε αυτό για τα θέματα τα εργασιακά. Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι έχουμε αναφορές για προβλήματα που υπάρχουν με το πώς τα κεφάλαια για την αηφόρο ανάπτυξη με το Περού και την Κολομβία έχουν εξελιχθεί. Και πρέπει να δούμε αν ε, υπάρχουν κάποιες ε, ε, υπερβάσεις ή παρεκκλήσεις από τη Συμφωνία Εμπορίου. Δεν θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα παρεκκλίνει από τις κατευθυντήριες γραμμές. Θα πρέπει λοιπόν να καλωσορίσουμε τα στοιχεία αυτά στην έκθεση που στοχεύουν στο να υπάρξει συμμόρφωση με αυτές τις αρχές. Και θα ήθελα να επικεντρωθούμε πολύ περισσότερο στη σχέση μας με τα κράτη της Λατινικής Αμερικής σε αυτά τα θέματα. Χαιρετίζω το θέμα του ότι καλό θα ήταν οι λατινοαμερικανικές χώρες να μπορέσουν να προαγάγουν τα θέματα, τα θεματολογικά αυτά ζητήματα στι σημερινή μας διατάξεις και καλωσορίζω αυτή την πρόταση στη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ θέλω να συγχαρώ τον εισηγητή για την έκθεση αυτή και φυσικά να εκφράσω και το ότι θα πρέπει επιτέλους να μπορέσουμε μέσω του ψηφίσματος να προχωρήσουμε και η, το, η σημερινός να ενταχθεί σε αυτή τη συμφωνία με την Κολομβία και το Περού και να μπορέσει έτσι και στη συνέχεια και να ενταχθεί και η Βολιβία. Όμως κάνουμε λόγο για μια συμφωνία. Είναι σημαντικό λοιπόν να μην ξεπερνάμε τα πλαίσια τα οποία έχουν τεθεί και να υπάρχει ένας συντονισμός με την κοινότητα, κράτη της κοινότητας ε, των Άνδεων. Είναι σημαντική η φόρος ανάπτυξη και για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα, αλλά ιδιαίτερα για το Εκουαδόρ. Και ως υπεύθυνη, μία από τις υπεύθυνες για αυτά τα θέματα σε αυτή την Κοινοβουλευτική Επιτροπή, δεν θα πρέπει μια και έχουμε εργαστεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα να μην αγνοήσουμε τη σπουδαιότητα αυτών των θεμάτων και ίσως θα υπάρξουν και τροπολογίες που θα κατατεθούν σχετικά. Παρακαλώ Μπορέλ στο τέλος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να προχωρήσουμε γρήγορα στην υπογραφή της έμβλογος συμφωνίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Σόλτς για την καλή δουλειά που έκανε και που μας υπενθύμησε τη σημασία που η οριστική συμφωνία θα έχει για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη βιώσιμη ανάπτυξη και για τα εργασιακά δικαιώματα. Συμφωνούμε από αυτών των θεμάτων 100%. Όμως μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα θέλαμε να τονίσουμε ότι τα δικά μας αιτήματα θα πρέπει να ακολουθούν την αρχή της ε, βαθμίας προσέγγισης και της θεματικής προτεραιότητας και να λάβουν υπόψη την ε, κοινωνικονομική κατάσταση της χώρας και τις ε, προσπάθειες που έχουν καταβληθεί όπως αναφέρονται στην επιστολή του Υπουργού του Εκουαδόρ. Γιατί πέρα από την εμπορική διάσταση της πτυχής της συμφωνίας, το θέμα είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την κοινωνία, το συνόλο και το πληθυσμό. Εμείς ως κοινοβούλιο και ως εκπρόσωποι των πολιτών θα πρέπει να διαρωτηθούμε στο πώς οι δικές μας προσπάθειες προωθούν τις αξίες τις οποίες πιστεύουμε και μπορούν να γίνουν η σωστή και αποτελεσματική απάντηση στη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτή η χώρα. Θα πρέπει επίσης να δώσουμε σημασία ούτω ώστε αυτές οι συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών να συνεισφέρουν μακροπρόθεσμα στην εξάλληψη των ισοτήτων και να μην χρησιμοποιηθούν από ισχυρά κέντρα όπου ως ε, μοχλούς για νέο απεικιοκρατισμό. Ε, μην ξεχνάμε ας πούμε τη μαζική αποδάσωση του Αμαζονίου. Όπω λέει ο Υπουργό στην επιγραφή του. Μην ξεχνάμε ότι και εμεί έχουμε ευθύνη και ολόκληρη η διεθνή κοινότητα. Η Ευρώπη θα πρέπει να είναι ένα μοντέλο ελπίδα και ευημερία για τη Λατινική Αμερική. Και είναι και για αυτού του πληθυσμού θα πρέπει να είναι, αλλά και για του πιο αδύναμου τα αδύναμα, του αδύναμους αυτή τη κοινωνία. Ε, τις αδυνάμες ομάδες, τις, τις γυναίκες κτλ. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε μία πιο διαφανή στάση, ε, να είναι πιο δραστήρια η Κομισιόν, θα πρέπει να λογοδοτήσει το Κοινοβούλιο για τη φάση υλοποίησης και εφαρμογή τη της συμφωνίας και ευχαριστούμε που το συζητάμε σήμερα αυτό το θέμα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Γιώργενσεν, επικεφαλής μονάδα στην Επιτροπή. Ευχαριστώ. Κάποια σύντομα σχόλια από πλευρά μου. Προφανώς καλωσορίζουμε την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου πρότασης ψηφίσματος που υποστηρίζει την ένταξη του σημερινού σε αυτή τη συμφωνία. Έχουμε εργαστεί υπέρ αυτού του αιτήματο κατά το παρελθόν σε σχέση με τις διαπραγματεύσεις. Θα ήθελα κάποια σύντομα σχόλια να κάνω σε κάποια στοιχεία αυτού του σχεδίου ψηφίσματος που δημιουργούν ίσως κάποιες ανησυχίες ε, για μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και απαιτούνται κάποιες αντιδράσεις, απαντήσεις από εμάς. Ε, βλέπουμε ότι εκφράζεται η άποψη του εισηγητή σε σχέση με την κατεύθυνση του σχεδίου ότι δεν υπάρχουν επαρκή μέτρα για την υλοποίηση των προγραμμάτων δράσης ε, της Κολομβίας και του Περού και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει ενημερωθεί επαρκώς. Εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ευθύς εξ αρχής κατανοήσαμε την σπουδαιότητα που δίνει στα δικαιώματα του ανθρώπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στα εργασιακά θέματα. Και όσο, όπως θα ενθυμίσετε, σαν, αντίδραση, σαν απάντηση της αντίδρασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεσμευθήκαμε να βοηθήσουμε, να επικουρήσουμε την Κολομβία και το Περού σχετικά και το κάναμε και δεσμευθήκαμε να χρησιμοποιήσουμε το πλαίσιο τα πλαίσια που καλύπτουν πολλά από τα θέματα που αφορούν αυτά τα έγγραφα, για παράδειγμα τα διάφορα κεφάλαια της συμφωνίας, αλλά επίσης και τα θέματα διαλόγου για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των ε, μέσων και μηχανισμών συνεργασίας. Το θέμα είναι κατά πόσο έχει επαρκώς ενημερωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από εμάς και έχουμε πολύ θετικές επιδόσεις εμείς σχετικά. Ενημερώσαμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για όλες αυτές ε, τις δραστηριότητες. Έχετε λάβει την έκθεση, ετήσια έκθεση υλοποίησης από πλευράς μας και, καθώς, ε, και για το αίτημα ενημέρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με τον Ιανουάριο 2014 και τον Ιανουάριο 2015 για την ε, ε, προώθηση των θεμάτων αυτών υπήρξε ενημέρωση κατά τον Μάρτιο 2014 για την Κολομβία και το Περού ενημερώσαμε τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και την Επιτροπή Ανάπτυξης και εσάς και αντιδράσαμε και σε ερωτήσεις τοποθετηθήκαμε σε ερωτήσεις ευρωβουλευτών Μία τελική παρατήρηση για το ε, εδάφιο, την παράγραφο 28 όπου ζητήθηκε σε σχέση με την, ε, το θεματολόγιο της υποεπιτροπής υπήρξε πλήρης ανταπόκριση και αν θα δείτε τις σημειώσεις που σας απεστάλησαν μετά τη συνάντηση που έγινε στη Μπογοτά στις 9 Ιουνίου σας διαθέσαμε πολύ υλικό και πάρα πολλά στοιχεία όπως ε, ζητήθηκε από πλευρά σας όλα τα θέματα της υποεπιτροπής καλύφθηκαν και προφανώς ε, είμαστε πρόθυμοι να συνεχίσουμε να διαθέτουμε αυτά τα στοιχεία και για το θεματολόγιο της Επιτροπής σας και της Υποεπιτροπής. Ευθυγραμμιζόμαστε απόλυτα λοιπόν με τα αιτήματά σας. Ευχαριστούμε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Εσείς τώρα παρακολουθείτε. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε αγαπητοί συνάδελφοι, εκπρόσωπε της Επιτροπής, Σίγουρα όλοι έχουν συνειδητοποιήσει ότι με το σχέδιο έκθεσης ή το σχέδιο ψηφίσματος ε, έχουμε κάποια σημεία που ε, συναπατίζουν μια απαιτητική μερίσια διάταξη όπου θέτουμε κέντρα βάρους ε, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει κέντρα βάρους για την επικύρωση αυτής της προσχώρησης και ταυτόχρονα Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι καλούμαστε να εμπλακούμε σε σχέση με τα επιμέρους σημεία και κάποιες εξειδικεύσεις απαιτούνται, κάποιες επισημάνσεις, κάποια αιτήματα που πρέπει να τύχουν συνέχειας και διευκρινήσεις σε σχέση με το σχέδιο ψηφίσματος που πρέπει συμπληρωματικά να ληφθούν υπόψη και καλούνται όλοι οι συνάδελφοι ενεργά να συμμετάσχουν από την Επιτροπή μας ιδιαίτερες και όδης εισηγητές. Τρία σύντομα σημεία στα, τα οποία αναφέρθηκαν στη συζήτηση. Πρόγραμμα δράσεων ή οδικός χάρτης. Βρισκόμαστε σε μια πολύ συγκεκριμένη ξεχωριστή συγκυρία ιστορικά. Εδώ και ένα έτος σχεδόν με τους Κολομβιανούς βρισκόμαστε σε άμεσες συζητήσεις, όμως Χωρίς οδικό χάρτη προσπαθήσαμε στο ψήφισμα να εντάξουμε κάποια στοιχεία που όμως καθορίζουν, δίνουν το πλαίσιο αυτών των στοιχείων για μια τέτοια συμφωνία και δείχνουν που υπάρχουν τα προτερήματα και τα πλεονεκτήματα κοινωνικά και οικονομικά για παράδειγμα όσον αφορά το Εκουαδόρ, τον Ισημερινό και που υπάρχουν κάποια άλλα σημεία τα οποία πρέπει να γίνουν σεβαστά και να εφαρμοστούν όσον αφορά τη διαδικασία προσχώρησης του Ισημερινού σε αυτή τη συμφωνία μια ξεχωριστή συγκυρία που καθιστά ίσως πιο περίπλοκη την κατάσταση για όλους τους εμπλεκόμενους και πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτή την ιδιομορφία. Δεύτερη παρατήρηση. Πιστεύω σίγουρα ότι πρέπει να συνειδητοποιήσουμε γιατί ο Ισημερινός μόνο το 2014 θέλει, ήθελε να προσχωρήσει σε αυτή τη συμφωνία υπάρχει μια ξεχωριστή οικονομική εξέλιξη στον Ισημερινό και μια απόφαση λοιπόν του επανεκλεγέντος Προέδρου και της κυβέρνησής του που δεν ήθελαν επί ένα χρονικό, συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να προσχωρήσουν σε αυτή τη συμφωνία, διότι οι εσωτερικοί όροι και προϋποθέσεις ήταν διαφορετικές και δεν είχαν αξιολογηθεί ως θετικοί και πρέπει αυτό να το λάβουμε ιδιαίτερα υπόψη και να λάβουμε υπόψη τα διαφορετικά συμφέροντα που ε, εμπνέουν το συμβαλόμενο αυτό μέρος ώστε να μπορεί να κινηθεί με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη λοιπόν η ξεχωριστή κατάσταση του εταίρου και να συνειδητοποιήσουμε αυτή την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Και αυτό απαιτεί επίσης μελλοντικά μια ε, ανοιχτή και ειλικρινή στο πλαίσιο της αντιμετώπιση εταίρων όταν έχουμε τέτοιου είδους εταιρικές συμφωνίες και σχέσεις που θα αποβαίνουν προς όφελος όλων των πολιτών, όλων των πολιτών στις ε, περιοχές και περιφέρειες του κόσμου με τις οποίες θα συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες και που πρέπει να αποβαίνουν προς όφελος αυτών. Επόμενη παρατήρηση. Σίγουρα τίθεται πάντα το θέμα ε, του γνώμονα. Με ποιο πύχη θα κρίνουμε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι σε σχέση με αυτά με αυτοπεποίθηση πρέπει να στραφούμε στο μέλλον και να δούμε από πού μπορούμε να αντλήσουμε πληροφορίες στρατηγικές για την υλοποίηση και να ονοματίσουμε, να απαριθμίσουμε με σαφή τρόπο αυτά τα στοιχεία ώστε οι πολίτες ε, ε, και στις δύο όχθες να γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται όταν συνάπτουμε τέτοιες συμφωνίες και να είναι πλήρης η ενημέρωση ώστε να μπορούμε να κατανοήσουμε γιατί συνάπτεται μια τέτοια συμφωνία σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή με συγκεκριμένους στόχους. Και στην περίπτωση του Ισημερινού είναι θέμα γενεάς που πρέπει να δικαιωθεί και να ε, προστατευτεί στην περιοχή για παράδειγμα η ζώνη του Αμαζονίου και των προβλημάτων που υπάρχουν εκεί. Γι' αυτό πρέπει με πολύ συγκεκριμένο τρόπο να λαμβάνουμε υπόψη τη βιοπικιλότητα και την προστασία της και το πώς μπορούν ο Ισημερινός και οι άλλα, τα άλλα γειτονικά κράτη της κοινότητας των άνδεων να μπορέσουν οικονομικά να αναπτυχθούν αλλά σεβόμενοι όλες αυτές τις πτυχές, το περιβάλλον και τη βιοπικιλότητα. Αδειμονώ να ακούσουμε το ποια συνέχεια θα τύχει πια συνέχεια στα τύχει αυτό το ψήφισμα και έτσι το έργο μας το οποίο επιτελέσαμε να μπορέσει να ευδοκιμήσει. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε θερμά. Πράγματι, η προθεσμία σε σχέση με την κατάθεση τροπολογιών είναι η 17η, 17η Ιουλίου. 12 το μεσημέρι. 12 το μεσημέρι. Και στις 21-22 Σεπτεμβρίου θα ψηφίσουμε μετά τις ε, σχετικές τροπολογίες. Θέλω να αναφέρω ότι σε σχέση με τις εμπορικές σχέσεις με τη Λατινική Αμερική θα έχουμε μια ακρόαση στις 19 Νοεμβρίου όπου σε ένα ευρύτερο πλαίσιο θα εξετάσουμε τα οικονομικά θέματα, οικονομικές σχέσεις, κοινωνικές σχέσεις κτλ. Σας ευχαριστώ θερμά. Περνάμε στο επόμενο σημείο, σημείο υπαριθμών 6 αγαπητοί συνάδελφοι. Πρόκειται για το θέμα της ε, σύμβασης για τη διαφάνεια όσον αφορά τις, ε, ε, τα θέματα επιδιαιτησίας και έχουμε εδώ κάτι το καινοφανές. Για πρώτη φορά στην συζήτηση έχουμε μία βιντεοδιάσκεψη την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Ήδη είχαμε μία ανταλλαγή με τον ε, Γενικό Γραμματέα Ουντσίπαλ υπό την αιγίδα ε, του οποίου του σώματος αυτού είχαμε τις διαδικασίες ISDS. Αυτή τη φορά ο Γενικός Γραμματέας δεν θα είναι προσωπικά παρόν, αλλά στην βίντεο διάσκεψη στο κέντρο θα μπορούμε να έχουμε επαφή μαζί του. Χαίρομαι λοιπόν που μπορούμε να τον δούμε σε, στην ε, μαγνητοσκόπηση. Ευχαριστώ θερμά για την υπομονή που είχε ώστε με αυτή τη διαδικασία με κάποια καθυστέρηση που είχαμε να μπορέσει να παρέμβει. Προτού του δώσω τον λόγο, θα δώσω σύντομα τον λόγο στον εισηγητή μας, ώστε για αυτή τη σύμβαση να μας πει δύο λόγια. Παρακαλώ εισηγητά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Όπως ακούσαμε τους τελευταίους μήνες, ξανά και ξανά, εδώ η Επιτροπή μας ε, συζητήσε με μεγάλο ζήλο, με μεγάλη συμμετοχή πολλών, τον, το θέμα της επίλυσης διαφορών μεταξύ κρατών και επενδυτών. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη στιγμή για να αντιμετωπίσουμε με επικοδομητικό τρόπο ε, ένα αυτό το θέμα με το Γενικό Γραμματέα της Ουσιτράλ τον οργανισμό που δημιουργήθηκε από τον ΟΗΕ για να προωθήσει την προοδευτική εναρμόνιση και ενοποίηση των κανόνων για το διεθνές εμπόριο. Το ψήφισμα ή μάλλον η επίλυση των διαφορών είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Ε, το Κοινοβούλιο το εξετάζει από τη σκοπιά της διαφάνειας. Διαφάνεια ε, στους κανόνες που διέπουν την ε, διαδικασία αυτή επίλυση διαφορών. Η μεγαλύτερη διαφάνεια είναι στόχος, γιατί μπορεί να εξασφαλίσει στους ενδιαφερόμενους του δημόσιου τομέα μεγαλύτερη γνώση για το πώς και πότε αποφασίζεται το θέμα αυτό στα πλαίσια της επίλυσης διαφορών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η επίλυση διαφορών μεταξύ κρατών και, ε, και και επενδύσεων μπορεί να αφορούν θέματα δημοσίου ενδιαφέροντος και συμφέροντος και μπορεί να επηρεάσουν και τα δημοσιονομικά μιας χώρας. Η δημοσιότητα, η διαφάνεια μας ε, διευκολύνει να καταλάβουμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε πιο ενιαίο τρόπο το δίκαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο μαζί με την, Επιτροπή, την αρμόδια Επιτροπή για το δίκαιο του ΟΗΕ προκειμένου να υπάρξουν ε, παγκόσμιοι κανόνε για τη διαφάνεια. Νομίζω ότι μια συνεργασία μεταξύ τη Φουνσιτράλ και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να ερμηνευτεί ω μια ευκαιρία για να διευκολύνουμε, να διευκολύνουμε και να ε, ενισχύσουμε το σύστημα επίλυσης διαφορών. Αυτή η διαφορά τι σημαίνει, ότι οποιαδήποτε διαφωνία ε, πολιτικής φύσεως, δικαιολογημένη, αιτιολογημένη, θα πρέπει να εξεταστεί, ούτως ώστε να βρούμε τον τρόπο για να διευκολύνουμε τη δυνατότητα συνεργασίας με αποφασιστικότητα. Γιατί ένα τέτοιο εργαλείο, υπενθυμίζουμε, ότι εκπροσωπεί, αφορά πάνω από 1.400 διμερείς συμφωνίες και θέλουμε αυτό το εργαλείο να γίνει πραγματικά εργαλείο διαφάνειας και πραγματικής δημοκρατίας. Νομίζω ότι πρέπει να αναφερθούμε σε μια ψηφοφορία που έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εδώ στην Επιτροπή μας μάλιστα για το θέμα αυτό του μηχανισμού επίλυσης διαφορών επενδυτών κράτους. Ε, και προσπαθήσαμε να δώσουμε μέσω της πληροφορία μας αυτής μια ισορροπημένη λύση, προς σωστή κατεύθυνση. Μια κατεύθυνση η οποία προωθήθηκε πολλές φορές από την Επιτροπή μας και από τα μέλη της Επιτροπής, αλλά και από την ίδια την Επίτροπο της Εσίλια Μάλστρομ. Μία άμεση έτσι, αντιπαράθεση, χωρίς ταμπού, χωρίς προκατασκευασμένες λύσεις, χωρίς ε, προαποφασισμένες επιλογές. Ο στόχος μας είναι να υλοποιήσουμε ένα κοινό στόχο. Να υπάρξει ένα εργαλείο το οποίο θα αναγνωρίζεται ως εργαλείο του διεθνούς ε, δικαίου και που θα επιτρέπει στο Κοινοβούλιο και θα επιτρέπει και στην Επιτροπή μας να προχωρήσει τον ε, προβληματισμό για την εμπορική πολιτική για να υιοθετηθούν πάντα οι καλύτερες δυνατές λύσεις. Οι αλλαγέ οι οποίε προωθήσαμε εδώ στην Επιτροπή νομίζω ότι πηγαίνουν προ αυτή κατεύθυνση. Δηλαδή, να προβλέπουμε ε, να υπάρχει μια δημόσια ακρόαση, να υπάρχει ένα ανεξάρτητος δικαστής και να υπάρχει και μια δυνατότητα έφεσης κατά των αποφάσεων. Διαφάνεια. Όταν μιλάμε για τη διαφάνεια, δεν πρέπει να θεωρήσουμε ότι αυτό είναι γράμμα κενό περιεχομένου το οποίο το χρησιμοποιούμε έτσι όπως να είναι, αλλά με συγκεκριμένο, μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Ε, και θα προχωρήσουμε σε αλλαγές, πρόσβαση σε έγγραφα, ε, δημόσια ακρόαση, τη δυνατότητα να παρουσιαστούν παρατηρήσεις, απόλυτη διαφάνεια στις αποφάσεις που θα λαμβάνονται. Επιφυλάσσομαι σε αυτή τη φάση. Θα κάνω ερωτήσεις και εγώ και στο γραμματέα και στην Επιτροπή. Ganz herzlichen Dank und... Σας ευχαριστούμε θερμά. Και έτσι τώρα στρεφόμαστε στη Βιέννη και πάμε στον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σοριόλ, και έχετε τον λόγο παρακαλώ. Good afternoon. Can you hear me? Καλό σας απόγευμα. Μπορείτε να με ακούσετε? Με ακούτε? Σας ευχαριστώ. Είναι χαρά να απευθύνομαι στην Κοινοβουλευτική σας Επιτροπή και σας ευχαριστώ που προσκαλέσετε την ε, Ansitral. Σε σχέση με το πλαίσιο αυτό για την, ε, τις δράσεις μας όσον αφορά την επιδιαιτησία όσον αφορά επενδυτές ε, και κράτη όχι μόνο για την Ευρώπη αλλά και παγκόσμιο εγχείρημα και παγκοσμίου ενδιαφέροντος και εμβέλειας σε πάμπολες επενδυτικές συμφωνίες. Ένας αυξημένος αριθμός, όλο και μεγαλύτερος αριθμός κρατών επανεξετάζουν τέτοιου είδους συμφωνίες επενδύσεων και οι πρόσφατες συμφωνίες λαμβάνουν υπόψη τις διατάξεις, τα δικαιώματα και υποχρεώσεις όσον αφορά τους επενδυτές και τα κράτη, καθώς επίσης και σε συνάφεια και συνεκτικότητα με άλλες πολιτικές ε, όσον αφορά την ανάπτυξη για παράδειγμα και την αηφόρο ανάπτυξη μεταξύ αυτών. Και υπάρχει και μία μετάθεση από τις ε, διμερείς τέτοιες συμφωνίες σε περιφερειακές συμφωνίες και αυτές έχουν ιδιαίτερες επιπτώσεις όσον αφορά τι επενδύσεις ε, και για την παγίωση των διατάξεων αυτών των πλαισίων ή και την αντιμετώπιση επικαλύψεων και την απλούστευση. Ας δώσω κάποιες πρώτες ενδείξεις ε, για το θέμα της διαφάνειας. Όπως γνωρίζουμε, η ANSITRAL είναι η επιτροπή που δημιουργήθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, την Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, με εντολή να εναρμονίσει και να εξυγχρονίσει αυτές τις διεθνείς συμφωνίες διεθνούς εμπορίου. Η σε σχέση με την δημιουργία σύγχρονων κανόνων που θα ρυθμίζει αυτές τις σχέσεις ε, σε ένα αντικειμενικό πλαίσιο μεταξύ κρατών και άλλων εμπλεκόμενων ώστε να υπάρχει η δυνατότητα εφαρμογής και ερμηνείας αυτών των διατάξεων. Ιδιαίτερα όσον αφορά την επιδιατησία, η Ansitral συνεισφέρει σημαντικά για την εκπόνηση και προαγωγή των διεθνών προδιαγραφών και διατάξεων. Η οικουμενική πρόσβαση στην ε, Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών όσον αφορά τις συμφωνίες αυτές είναι ένα παράδειγμα. Η επιτυχία της Σύμβασης της Νέας Υόρκης ε, και των μέσων της ε, συνεισφέρουν στον ρόλο της επιδιαιτησίας ως ένα ειρηνικό μέσο για τη διευθέτηση των ε, τριβών, διεθνών προβλημάτων και ε, διαφορών καθώς επίσης και μια διαιτησία που θα βασίζεται στις διατάξεις της Ανσιτράλ όσον αφορά το πλαίσιο το οποίο κατά το 1995 δημιουργήθηκε καθώς επίσης και την εφαρμογή των κανόνων αυτών που από το 1976 θεσπίστηκαν. Εργαζόμενοι με συνέπεια σε σχέση με την αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων θέλω να σας ενημερώσω για το πρόσφατο έργο για τη διαφάνεια της Ancitral που εξελίχθηκε σε σχέση με την προηγούμενη πείρα μας. Μία από τις ανησυχίες που εκφράζεται σε σχέση με τις επενδύσεις είναι ότι οι συναφείς διαδικασίες και τα αποτελέσματα έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα και δεν αποκαλύπτονται ακόμα και όταν ε, τα θέματα αυτά αφορούν κρατικά συμφέροντα. Αυτά τα θέματα δημιουργούν ανησυχίες ε, και πρέπει να αντιμετωπιστούν. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο το έργο της Άνσιτρά, για την διαφάνεια όσον αφορά την επιδιαιτησία τον Οκτώβριο 2010 και μετά από τρία έτη εργασιών το 2013 οι κανόνες και κανονισμοί για την διαφάνεια οι οποίοι θα λαμβάνονται υπόψη όσον αφορά τις σχέσεις επενδυτών και κρατών που υιοθετήθηκαν και που συναποτελούν μια σημαντική αλλαγή από το status quo όσον αφορά τις προηγούμενες ε, διαδικασίες επιδιατησίας που ε, λάμβαναν χώρα και κλεισμένων των θυρών ακόμα και αν τύχανε ιδιαίτερης προσοχής ε, από πλευράς των μέσων τέτοιου είδους υποθέσεις χωρίς να υπησέλθω σε λεπτομέρειες οι κανόνες δίνουν ένα διαδικαστικό πλαίσιο που δίνει στο κοινό μια ευρύτερη πρόσβαση όσον αφορά τα έγγραφα και τα στοιχεία αυτά σε σχέση με αυτά τα θέματα. Οι κανόνες και κανονισμοί προβλέπουν ανοιχτών θυρών διαπραγματεύσεις, δημόσιες διαπραγματεύσεις και την δυνατότητα τρίτων μερών να υποβάλουν προτάσεις. Συμπεριλαμβάνουν αξιόπιστες διατάξεις ε, για την διαφύλαξη σημαντικών πληροφοριών. Και το πιο σημαντικό είναι προσπαθούν να εξισορροπήσουν το δημόσιο συμφέρον όσον αφορά τις πληροφορίες και τα συμφέροντα εμπλεκομένων μερών ώστε να υπάρχει μια ε, δίκαια ε, αντιμετώπιση των συμφερόντων τους. Η υιοθέτηση των κανόνων διαφάνειας όσον αφορά ε, το πλαίσιο διαφάνειας για τέτοιου είδους συμφωνίες έχουν δώσει την δυνατότητα μιας τέτοιας σύμβασης ε, που είναι δυνατόν να εμπλέκει όλους τους οργανισμούς εκείνους ε, που επιθυμούν να καταστήσουν εφαρμοστέους τους κανονισμούς ε, αυτούς σε σχέση με τις δικές τους συμφωνίες και συνθήκες και να μπορέσουν έτσι να λειτουργήσουν από το 2014 στην Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών που ενέκρινε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την διαφάνεια όσον αφορά τις συμβάσεις και συνθήκες για τις σχέσεις επενδυτών και κρατών. Και η σύμβαση αυτή συμπεριλήφθηκε ιδιαίτερα με την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτό το ευρύτερο πλαίσιο. Σαν συνέπεια τούτου συμπληρώνεται το υφιστάμενο πλαίσιο συνθήκων σε σχέση με τις υποχρεώσεις ε, που διέπουν τους εμπλεκόμενους. Σε σχέση με όσους ε, συμμετέχουν σε μια περιφερειακή οργάνωση και εκφράζουν την ε, ανάγκη να ισχύουν οι διατάξεις διαφάνειας όσον αφορά τις επενδύσεις μέσα σε αυτά τα πλαίσια. Επίσης ε, παρέχεται η ελαστικότητα, η ευληγησία, ώστε να μπορούν τα εμπλεκόμενα μέρη να εκφράζουν τις επιφυλάξεις τους ε, σε σχέση με τις διατάξεις αυτές, ιδιαίτερα όσον αφορά συνθήκες επενδύσεων ή συγκεκριμένους κανόνες και κανονισμούς. <clears throat> Η συνθήκη αυτή για το Πορλουί, Πορλουί του Μαυρικίου Κατά τις 17 ε, Μαρτίου 2015 ξεκίνησε η διαδικασία επικύρωσης και ε, στα κεντρικά γραφεία της ε, Νέας Υόρκης βρίσκεται υπό εξέλιξη αυτή η προσέγγιση. Έχουμε και έναν αριθμό ευρωπαϊκών κρατών, Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία καθώς επίσης και τον Καναδά από την άλλη πλευρά και τη ΣΥΠΑ που συμμετέχουν. Οι κανόνες για τη διαφάνεια που προβλέπονται σε σχέση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών που έχει ε, και την αρμοδιότητα ε, λειτουργίας ενός μητρώου για τις διατάξεις αυτές και οι πληροφορίες ε, είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα του μέσου και υπάρχει η πρόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να υποστηρίξει την λειτουργία του Μητρώου Διαφάνειας για την οποία αυτή η δράση έχει εκφραστεί η πρόθεσή τους. Οι κανόνες ε, διαφάνειας σε σχέση με τη συνθήκη και το Μητρώο Διαφάνειας είναι τα πρόσφατα αποτελέσματα λοιπόν μιας πολυμερούς προσπάθειας για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσον αφορά τα θέματα επιδιαιτησίας ε, επενδυτών και κρατών, λαμβάνοντας υπόψη και το δημόσιο συμφέρον αλλά επίσης και το ιδιωτικό συμφέρον των εμπλεκόμενων για την επίλυση τέτοιου είδους διαφορών με έναν δίκαιο ε, τρόπο. Και επίσης ε, συνεισφέρουμε σε ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την λειτουργία αυτών των διατάξεων όσον αφορά τα διεθνή θέματα τα διεθνή επενδυτικά θέματα. Επίσης, οι διατάξεις για τη διαφάνεια θα συνεισφέρουν σημαντικά για την διεύρυνση της διαφάνειας όσον αφορά την επίλυση αυτών των θεμάτων μέσα από αυτό το καθεστώς και θα πρέπει η διαφάνεια έτσι να κατανοείται μέσα στο πλαίσιο των άμεσων αλλοδαπών ε, ε, επενδύσεων ως ένα μέσο για την αηφορία. Έχοντας στη διάθεσή μας ε, τα στοιχεία τα οποία μας ενδιαφέρουν για τέτοιου είδους δράσεις, συνεισφέρουμε στο να υπάρχει ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης για την λειτουργία τέτοιου είδους δράσεων και επιπλέον ε, ένα σημαντικό βήμα για να ανταποκριθούμε στις ε, αυξημένες προκλήσεις όσον αφορά την νομιμότητα, όσον αφορά το διεθνές δίκαιο για τις επενδύσεις ε, και την επιδιαιτησία. Τα θέματα διαφάνειας διευρύνουν την κατανόηση των πολιτών για τα θέματα επιδιαιτησίας και αυξάνουν και το επίπεδο αξιοπιστίας συνολικά. Οι παρατηρήσεις για τις μεταρρυθμίσεις σε σχέση με αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να τονίσω σήμερα ότι το έργο που επιτελείται από την Ancitral <clears throat> κανονικά αυξάνει την διαφάνεια και μπορεί να προλιάνει το έδαφος ώστε να υπάρχει ανταπόκριση για ακόμα μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις και συνεισφορά για τον εξυγχρονισμό συνολικά του συνολικού πλαισίου για τις επενδύσεις και πρέπει να κατανοήσουμε ότι υπάρχουν πάνω από 3.000 ε, συμβάσεις ε, επενδύσεων παγκόσμια ένα τεράστιο ποσοστό σε σχέση με αυτές ε, τις συμβάσεις βρίσκονται υπό, υπό την αιγίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένας μηχανισμός ώστε να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις. Και εξετάζουμε λοιπόν τη δυνατότητα να μπορέσουμε να εμπλακούμε σε σχέση με αυτές τις ε, προτάσεις. Η μεταρρύθμιση θα πρέπει να, λαμβάνει, να λαμβάνουν υπόψη τις, ε, τους διαφορετικούς όρους αυτών των πλαισίων. Ωστόσο δεν είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Ένωση ή τα κράτη-μέλη μόνα τους μπορούν να αντιμετωπίσουν μεμονωμένα. <clears throat> Μια ευρωπαϊκή προσέγγιση χωρίς την συμφωνία των εταίρων εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα οδηγήσει σε μια ημιτελή κατάσταση πραγμάτων. Και γι' αυτό υιοθετώντα την προσέγγιση, ε, πολυμερή προσέγγιση για την διαφάνεια, για την δημιουργία ενός μηχανισμού όπως αυτής της σύμβασης, θα πρέπει να μπορέσουμε να προχωρήσουμε πιο αποτελεσματικά. Και έτσι λαμβάνει την ε, μορφή μιας ε, αμφίδρομης δράσης λαμβάνοντας υπόψη τις υφιστάμενες συμφωνίες διότι υπάρχει εδώ η τάση υπέρ της διαφάνειας σε σχέση με ε, την διαφάνεια των επενδύσεων είναι κάτι σχετικά ε, πρόσφατο. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούμε να τα λάβουμε υπόψη μας κατά την προετοιμασία μιας σύμβασης. Αλλά όταν επεκταθούμε σε δικονομικά θέματα, αυτό ε, πρέπει να το δούμε, ε, δηλαδή στις ισχύουσες επενδυτικές συμφωνίες, αυτό θα πρέπει να το δούμε. Και πρέπει να το εξετάσουμε πάρα πολύ προσεκτικά. Σε ό,τι αφορά την... Επειδή υπάρχουν πάρα πολλές ε, λεπτομέρειες ε, στη δομή των επενδυτικών συμφωνιών και επειδή υπάρχει και δημόσια προσοχή που δίδεται τελευταία σε αυτά τα θέματα, το πιο σημαντικό στοιχείο είναι η πολιτική θέληση των εμπλεκόμενων για να φτάσουν σε συνένεση επί της ουσίας μόνο όταν και εφόσον αυτό επιτευχθεί, και ελπίζουμε ότι θα γίνει με τους κανόνες περί διαφάνειας, ένας παρόμοιος μηχανισμός με τη σύμβαση περί θα μπορούσε να εξεταστεί. Ας κάνουμε προτάσεις, Φερρυπίν, για να δημιουργήσουμε ένα μηχανισμό ε, τύπου επενδυτικό δικαστήριο. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να εφαρμόσουμε μια τέτοια μεταρρύθμιση θα μπορούσαμε να το συμπεριλάβουμε σε μία από τις καινούργιες επενδυτικές ή εμπορικές συμφωνίες, ας πούμε. Αυτό όμως θα είχε μηδαμινή επίπτωση στην ε, διαιτησία ε, και σε συμφωνίες ε, που έχουμε ήδη και που είναι πολύ άριθμες. Μία άλλη προσέγγιση θα μπορούσε να ήταν να δημιουργήσουμε ένα χωριστό φορέα που θα έχει το καθήκον να, και την ευθύνη να χρησιμοποιεί τους σημερινούς, τους ισχύοντες μηχανισμούς, που θα πρέπει όμως ε, να τροποποιηθούν αναλα... αναλόγως. Ούτως ή άλλως θα χρειαστεί πάρα πολύς χρόνος και προσπάθεια για να φτάσουμε σε συμφωνία επί της ουσίας. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει ανάγκη για ένα τέτοιον επιπρόσθετο μηχανισμό. Και επίσης θα πρέπει να επιλέξουμε την κατάλληλη προσέγγιση. Ίσως πιο προβληματικό θα ήταν ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φόρουμ για μια τέτοια ενδελεχή συζήτηση. Οι συζητήσεις που γίνονται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ε, γίνονται κατακαιρματισμένα σε πολλιά αριθμούς διεθνείς και πολυμερείς οργανισμούς και αφορούν διάφορα θέματα. Με... Και οι συζητήσεις είναι πάρα πολύ γενικόλογες. Οποιαδήποτε συγκεκριμένη διαδικασία μεταρρύθμισης απαιτεί ένα πραγματικό φόρουμ όπου τα κράτη οι περιφερικές ε, οικονομικές ε, οργανώσεις όπως η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και φορείς διαιτησίας το δικαστήριο διαιτησίας, ε, εμπορικά επιμελητήρια και άλλοι εμπορευόμενοι όπως ακαδημαϊκοί, άνθρωποι που ασχολούνται με τα θέματα αυτά, διάφορες οργανώσεις μπορούν να βρεθούν μαζί και να ανταλλάξουν απόψεις. Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα και πιστεύω Εκεί η Αντσιτράλ μπορεί να συνεισφέρει στην διαδικασία, όπως φαίνεται και από τη δουλειά που έχει κάνει για τη διαφάνεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και με μεγάλη χαρά θα ακούσω και θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συνοπτική παρέμβαση. Υπάρχουν συγκεκριμένα ερωτήματα ο κύριος Σίκα, ο κύριος Ζάρντι, ο Σάρκε και ο κύριος Σόλτς. Συγκεκριμένα όμως ερωτήματα δεν έχουμε πολύ χρόνο. Σίκαου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Ανσιτράλ γιατί μας εξήγησε και μας είπε πράγματα πολύ ενδιαφέροντα Ποια αξιολόγηση κάνει η Ανσιτράλ για τον μηχανισμό ISDS, τον μηχανισμό επίλυση διαφορών ε, επενδυτή κράτου, λαμβάνοντα υπόψη τι τελευταίε προτάσει τη Επιτρόπου Μάλτσομ και του προσανατολισμού ε, που δώσαμε μέσω τη ψηφοφορία επί του ψηφίσματο στο Κοινοβούλιο του κυρίου Σανταλούνες που δεν είναι παρόν αλλά μου ζήτησε να θέσω ερωτήματα όχι προς τον προσκεκλημένο μας τον οποίο ευχαριστώ αλλά προς την Κομισιόν μάλλον δεν ξέρω αν είναι ο καταλληλότερος χρόνος και τόπος εδώ θα προσπαθήσω όμως γιατί και εγώ πρέπει να φύγω και οι βοηθοί μου θα καταγράψουν τις απαντήσεις. Σε τι, χρονοδιά, χρονοδιάγραμμα προβλέπει η Κομισιόν για τη συμφωνία με το Συμβούλιο ως προς το θέμα. Κάτι γρήγορο ή κάτι που θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Δεύτερο ερώτημα. Τι επικάλυψη βλέπει η Κομισιόν με τη συμφωνία της Συγκαπούρης, με την υποβολή του αιτήματος της διασία της Συγκαπούρης στο δικαστήριο ως προς την συμφωνία ε, της συνθήκης Λισαβόνας Τρίτων μπορεί μέχρι το τέλος του χρόνου να συμφωνηθεί και για την Ανσιτράλ τελικά πώς μπορεί να δημιουργηθεί ένα διεθνές δικαστήριο επενδύσεων. Ευχαριστώ η Μάρικη. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και για την πρωτότυπη αυτή τηλεδιάσκεψη από την UNCTRAL στα Έθνη, των Ηνωμένων Εθνών. Είναι σημαντικό για μας να τονίσουμε την πολυπλευρικότητα του συστήματος ακόμη κι αν για την προστασία των επενδύσεων φαίνεται ότι τονίζουμε μάλλον το TTIP στη συζήτηση μας αυτή τη στιγμή. Ο λόγος για τον οποίο βρίσκω ότι είναι σημαντική η σημερινή συζήτηση και ο ρόλος των ΗΠΑ είναι γιατί θα ήταν προφανώς λάθος να περιοριστούμε μόνο στο TTIP στις συζήτηση μας και το ISDS. Αλλά αυτό δυστυχώς συμβαίνει. Καταλαβαίνω γιατί πολιτικά είναι τόσο ελκυστικό, αλλά δεν λύνει τις δικές μου τουλάχιστον ευρύτερες ανησυχίες, ιδιαίτερα ως προς τα, τις υπάρχουσες περίπου 1400 συμφωνίες, εμπορικές συμφωνίες που περιέχουν και ρήτρες ε, για τις επενδύσεις και την προστασία τους. Αυτό λοιπόν μάλλον κάτι που αφορά όλους εμάς και την ευθύνη μας εδώ στην Ευρώπη. Δεν ξέρω αν είναι σωστές οι πληροφορίες μου, αλλά νομίζω ότι τον Ιανουάριο η Κομισιόν ανέλαβε την πρωτοβουλία να αναλάβει περισσότερες ε, πρωτοβουλίες διαφάνειας for greater access μεταξύ των οποίων και πρόσβαση στα έγγραφα. Έγινε εδώ μια πολύ ζωηρή συζήτηση στην Ένωση και το Κοινοβούλιο έπαιξε ρόλο και η Κομισιόν αλλά και οι Αμερικανοί συναδελφοί μας που ζητούσαν όλοι μαζί πρόσβαση στην πληροφόρηση. Αλλά άλλη είναι η τάση που ισχύει στα κράτη-μέλη. Αν λοιπόν οι σωστές πληροφορίες μόνο έξι χώρες μέλη υπέγραψαν αυτή την πρωτοβουλία διαφάνεια. Σωστό είναι αυτό. Αν ο κύριος από τη Βιέννη μπορεί να μας το επιβεβαιώσει. Πάντως φαίνεται πολύ χαμηλός ο αριθμός, αν και μπορεί να με, από τότε με δύο-τρεις χώρες παραπάνω να έχουν υπογράψει. Αλλά δεν συμβαδίζει καθόλου με τις προσπάθειες και τις σκέψεις που αναλύουμε εμείς εδώ. Θα ήθελα να μάθω πόσα κράτη-μέλη τελικά υπέγραψαν αυτή την πρωτοβουλία ή προσπάθεια διαφάνειας. Χέλμουτ Σόλτς. Ευχαριστώ και εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα για το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι σήμερα αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα και συμφωνούμε για την ε, σύμβαση για τη διαφάνεια και για την επιδιαιτησία. Υπάρχουν κάποια κενά ακόμα και κάποιες ε, ρογμές που πρέπει να ε, κλείσουν για να αποφύγουμε την διήθηση πληροφοριών όσον αφορά τέτοιου είδους ε, ε, διαφορές και είναι ένα σημαντικό θέμα και πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο για να μπορούμε να είμαστε πιο αποτελεσματικοί να λάβουμε υπόψη σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση αυτά τα ζητήματα αποτελούμε συμβαλόμενο μέρος σε αυτή τη σύμβαση. Τι σημαίνει λοιπόν για σας αυτό όσον αφορά τις ευθύνες για το διεθνές εμπόριο και την επενδυτική πολιτική σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σημαίνει ότι η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συναποτελεί τμήμα αυτής της σύμβασης μήπως. Ε, τότε θα πρέπει να κάνουμε τα του οίκου μας, το έργο μας, τη δουλειά μας σωστά και να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη επιτέλους να προσχωρήσουν και να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο είναι μίζωνο σημασία ε, θέμα. Όταν έχουμε συμφωνίες όπως την TTIP ε, ε, και θέλουμε να δημιουργηθεί κάτι όπως ένας διεθνής μηχανισμός ή ένα διεθνές σώμα μετά από μια περίοδο διαβούλευσης, πώς θεωρείτε εσείς το θέμα αυτό για τη διαφάνεια. Επειδή για παράδειγμα οι επενδυτές συνεπάγονται ε, ένα μεγάλο ποσοστό αυτών των ε, κονδυλίων ε, και της δράσης των κρατών. Υπάρχει κάποια αντιστάθμιση Προς αυτή την κατεύθυνση βαίνει το ερώτημά μου. Ίσως θα μπορούσατε να προσθέσετε κάποιες πρόσθετες πληροφορίες λοιπόν στα όσα αναφέρατε. Ευχαριστώ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρέμβει. Πράγματι <clears throat> εκκλείσει βάση το άρθρο 207 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δικαίωμα να εντάσσεται και να προσυπογράφει ε, τέτοιου είδους συμβάσεις. Και τώρα υπάρχει τροχοπέδηση από τα κράτη-μέλη. Λοιπόν, εσείς σου έχετε τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που θα ήθελα να πω, αλλά λόγω χρόνου θα είμαι λακωνικός και θα επικεντρωθώ στα θέματα τα οποία προέκυψαν από την ανταλλαγή. Είναι μια πολύ σημαντική σύμβαση, γιατί είναι η πρώτη επιτυχή σύμβαση που μεταρρυθμίζει μία, το διεθνές επενδυτικό δίκαιο και την διεθνή επενδυτική πολιτική. Γι' αυτό ακριβώ το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική σύμβαση αυτή. Η Κομισιόν, όπω είπατε, έκανε μια πρόταση για την υπογραφή αυτή τη συμφωνία τον Ιανουάριο του 2015. Αυτή η απόφαση συμπεριλαμβάνει και την υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την εξοδότηση από τα κράτη-μέλη. Έχει να κάνει με το θέμα των αρμοδιοτήτων. Ε, την εξοδότηση από τα κράτη-μέλη. Η απόφαση δεν έχει αυτηθεί ακόμα. Ήταν αδύνατο να βρεθεί συνένεση στο Συμβούλιο για να υιοθετηθεί η απόφαση αυτή. Η Κομισιόν ελπίζει ότι μπορούμε να προχωρήσουμε γρήγορα για... και για να απαντήσω σε μία από τις ερωτήσεις ε, που τέθηκαν χάρη στην Λουξεμβουργιαζική Προεδρία και να υιοθετηθεί η αλλά πρέπει να το δούμε αυτό αν θα γίνει έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσυπογράψει τη συνθήκη αυτή που είναι η μοναδική ε, συνθήκη που είμαστε μέλη και, τα κράτη-μέλη να προσυπογράψουν, ώστε να την εφαρμόσουν στις 1.400 αυτές ε, ισχύουσες συνθήκες προσυπογράψουν και να την εφαρμόσουν σε αυτές τις συνθήκες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα προσυπογράψει ως τμήμα του γενικού κινήματος που υπάρχει για τη μεταρρύθμιση του διεθνούς επενδυτικού καθεστώτος. Γιατί αυτό το σύστημα είναι ένα σύστημα που προσπαθεί να εφαρμόσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στα διαδικαστικά θέματα του επενδυτικού καθεστώτος. Ο κύριος Σόντερ Λούνς έκανε μια ερώτηση. Δεν συνδέεται άμεσα με το δικαστήριο της Σιγκαπούρης αυτό. Υπάρχουν κάποια θέματα λεπτά, όπως ξέρουμε, που έχει να κάνει, έχουν να κάνουν με τα θέματα των αρμοδιοτήτων. Αλλά δεν συνδέεται άμεσα με το δικαστήριο αυτό της Σιγκαπούρης. Συγγνώμη, είναι την υπόθεση της Σιγκαπούρης. Εμείς θέλουμε να περάσει το θέμα τώρα αυτό από το Συμβούλιο σύντομα, ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του όπως προβλέπετε, ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπογράψει και να επικυρώσει τη συμφωνία συνεχεία. Θέλουμε να προχωρήσουμε λοιπόν πολύ σύντομα και ελπίζουμε ότι θα επανέλθουμε στην Επιτροπή σας ε, με τελικά αποτελέσματα σύντομα. Ο Γενικός Γραμματέας τώρα θα ήθελα να απαντήσει σύντομα στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Και εγώ θα είμαι όσο πιο λακωνικός γίνεται. Καταρχάς, έγινε μια ερώτηση για τα στοιχεία. Για το πόσες υπογραφές έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έξι, νομίζω, είναι το σωστό νούμερο. Αυτή τη στιγμή έξι κράτη-μέλη. Εμείς δεν μπορούμε να σας πούμε πώς θα προχωρήσετε. Φυσικά, εμείς κάνουμε έκκληση, θερμή έκκληση να προσέξετε αυτή τη σύμβαση, γιατί αξίζει να την προσέξετε και να την λάβετε υπόψη σας. Ξέρουμε ότι πάντα χρειάζεται χρόνος, ούτως ώστε αυτά τα κείμενα του εμπορικού δικαίου να επικυρωθούν, να υπογραφούν καταρχά και να επικυρωθούν με συνεχεία. Όσο πιο νωρίς ξεκινήσουμε, τόσο το καλύτερο. Κάποιος είπε ότι πρέπει να γίνουν διάφορα πράγματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό είναι αυτό που λέτε, που ακούγεται και ελπίζουμε και τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεπεράσουν τις δυσκολίες ή τις αβεβαιότητες. Τονίζω ξανά και ξανά τη σημασία που έχει η δράση των Ευρωπαϊκών κρατών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως περιφερειακό θεσμικό όργανο. Γιατί περιμένουν το μήνυμα που θα στείλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το συνόλου στον υπόλοιπο κόσμο. Ε, το ερώτημα που τέθηκε, αρκεί η διαφάνεια, όχι προφανώς. Και πώς αυτό αλληλεπιδρά με το project για να δημιουργήσουμε ένα επενδυτικό δικαστήριο. Είναι πολύ νωρί να σχολιάσουμε λεπτομερώς το σχέδιο αυτό δημιουργίας Ευρωπαϊκού ή Διεθνούς Επενδυτικού Δικαστηρίου. Αυτό που είναι μάλλον σίγουρο σε αυτή τη φάση είναι ότι αυτό το project, αν προχωρήσει, αυτό το σχέδιο προχωρήσει, θα είναι μια μακρά και περίπλοκη διαδικασία και θα εγείρει ενδιαφέροντα και δύσκολα προβλήματα συμβατότητας και σεβασμού των προϋπαρχουσών συμφωνιών και συνθήκων. Επομένως, το, η θέση μας, Πρόεδρε, είναι ότι εξετάζουμε το θέμα αυτό με μεγάλο ενδιαφέρον και οτιδήποτε και αν συμβεί με το σχέδιο αυτό δημιουργία διεθνούς δικαστηρίου, διεθνούς δικαστηρίου διατησίας το ισχύον σύστημα θα πρέπει να βελτιωθεί ούτως ή άλλως, να μεταρρυθμιστεί ούτως ώστε να λειτουργεί πιο καλά, όσο καλύτερα μπορούμε και το, η προσπάθεια διαφάνειας, το σχέδιο αυτό διαφάνειας ήταν το πρώτο βήμα. Αλλά δεν είναι το μοναδικό και τελευταίο βήμα. Τώρα, τις τελευταίες μέρες, στην σύνοδο, την ετήσια σύνοδο που κάνουμε στη Βιέννα, λάβαμε την εντολή να προχωρήσουμε και να συζητήσουμε θέματα που αφορούν ένα πιθανό κώδικα διοντολογίας και διαιτητές, για τους διαιτητές, και το δέμα του, διαιτητών θα πρέπει να το δούμε ή μάλλον οι διαιτητές θα πρέπει να το δουν αυτό το θέμα λεπτομερώς, σε ό,τι αφορά το μηχανισμό ε, προσφυγών. Σίγουρα θα πρέπει να κάνουμε μια ενδελεχή έρευνα και μελέτη των τεχνικών πτυχών ενός τέτοιου μηχανισμού προσφυγών σε σχέση με τις ισχύουσες δομές που αφορούν την ε, σύμβαση της Νέας Υόρκης και την σύμβαση του 1965. Δεν είμαι σίγουρος ότι όλες οι επιπτώσεις ε, δημιουργίας ενός ε, μηχανισμού προσφυγών ε, έχουν αναλυθεί πλήρως. Ειδικά σε σχέση με τη σύμβαση της Νέας Υόρκης. Δεν έχουμε ακόμα λάβει εντολή να εξετάσουμε κάτι τέτοιο και σίγουρα είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια στιγμή εάν θέλουμε το ισχύον σύστημα να διορθωθεί και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του. Όλα αυτά, Πρόεδρε, φυσικά γίνονται με την επιφύλαξη του τι μπορεί να συμβεί στον τομέα της δημιουργίας αυτού του νέου θεσμού. Του δικαστηρίου δηλαδή αυτού. Όλα αυτά τα παρακολουθήσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και κλείνοντας θα ήθελα να σας πω ότι η Άνση είναι ένα φόρουμ το οποίο χάρη στη δουλειά που έχει κάνει για ε, θέματα εμπορικής διατησίας έχει αποκτήσει φήμη και μόνο πρόσφατα συνειδητοποίησε την επίπτωση που έχει δουλειά της στον τομέα των διατησιών για θέματα επενδύσεων. Ε, και είναι σημαντικό αυτό σε σχέση με το μηχανισμό ISDS, Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών Επενδυτή Κράτους. Αλλά εδώ θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, θα συνεχίσουμε την έρευνα όσο καλύτερα μπορούμε και αν μας δοθούν οι κατάλληλες ε, εντολές από τα κράτη, θα κάνουμε και την κατάλληλη προετοιμασία και δουλειά. Ευχαριστούμε. Ο εισηγητής μας, ο κύριος Σάικο. Ο κύριος Σάικο. Ευχαριστώ το Γενικό Γραμματέα για την ευκαιρία που μας έδωσε να μιλήσουμε για αυτό το θέμα και τους συναδέλφους που με τη συνεισφορά τους ε, βοήθησαν και αυτοί στην, στην υπάρξει προβληματισμός για αυτά τα θέματα. Είναι περίπλοκο το θέμα. Έχουμε την ευκαιρία να πούμε ότι ο αριθμός των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσυπέγραψαν τη σύμβαση ε, τελικά θα αυξηθεί και καλό και την Λουξεμβουργέζικη Προεδρία να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, ούτω ώστε να βοηθήσουμε και εμείς ε, στην εφαρμογή των ε, διατάξεων της Σύμβασης Αντσιτράλ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Γραμματεύ για τη διαθεσιμότητά σας και γιατί μας δείξατε, δώσατε μερικές από τις απόψεις σας για τη δουλειά σας. Ευχαριστώ και τους τεχνικούς που πραγματοποίησαν αυτή την καταπληκτική τηλεδιάσκεψη που γίνεται για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας. Ευχαριστούμε λοιπόν τη Βιέννη και όλους. Τελειώνει αυτό το σημείο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.